Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η προηγουμένη συνεδρία των συντονιστών. Έλαβε δε υπόψη τις ανακοινώσεις ε, της ε, Προέδρου. Να σας πω λοιπόν τι συζητήσαμε. Την 10η Απριλίου έχει επιβεβαιωθεί η ακρόαση για την πρωτοβουλία των πολιτών ένας από εμά, ο Άνω Βάς, ε, έχει μοιραστεί στα μέλη της Επιτροπής το πρόγραμμα αυτής της ε, ακρόασης της 10ης Απριλίου να σας πω ότι είναι η δεύτερη ακρόαση μετά από την πρωτοβουλία των πολιτών ε, για το νερό ε, και ολοκληρώνεται και αυτή πριν από την ολοκλήρωση της ε, θητείας, πριν από το τέλος της θητείας. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει να εκπροσωπηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ε, για τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικέ ανάγκες ε, βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 ε, και είπαμε επίσης ότι στη θεσμική ομάδα που θα εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο σε αυτήν την διάσκεψη θα συμμετάσχουμε και εμείς μαζί με εκπροσώπους της Επιτροπής Ελευθεριών των Πολιτών και Απασχόλησης. Επίσης, είπαμε ότι παρότι ε, θα έχει ολοκληρωθεί ας πούμε η θητεία ε, του παρόντος κοινοβουλίου ε, αλλά δεν θα έχει ξεκινήσει ακόμα η πραγματική λειτουργία της επόμενης θα στείλουμε αντιπρόσωπο της γραμματείας στο ένα το περιφερειακό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των, των Διάμεσολαβητών που θα λάβει χώρα στην Ουαλία, στο Κάρδιφ από 22 μέχρι 24 Ιουνίου του 2004 2014. Το ίδιο θα συμβεί και στην ε, συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου ε, των Διαμεσολαβητών. Ε, το σεμινάριο αυτό θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο από 27-29 Απριλίου. Εάν και εφόσον υπάρχουν μέλη της Επιτροπής τα οποία έχουν διάθεση και πρόθεση να συμμετάσχουν σε αυτό το σεμινάριο, παρακαλώ να μας το πούν. Επίσης είπαμε ότι έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία σχετικά σχετικά με τις αναφορές οι οποίες έχουν υποβληθεί έχουν γίνει συνόψεις και σας έχουν διανεμηθεί μέχρι το 1375 κάθετος 2013 και Επίσης να πούμε ότι λάβαμε μια θετική και ιδιαίτερως ενθαρρυντική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Προεδρία, ε, από την Ελληνική συγγνώμη, Προεδρία ε, όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση και το πολιτικό άσυλο. Ε, δεν έχω τίποτα άλλο ή μάλλον όχι. Να σας πω ότι οι συντονιστές αποφάσισαν ε, για την αναφορά που είχε εγγραφεί στο σημείο 13 της ημερησίας διατάξεως να ζητήσουν μελέτη από το τμήμα μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε συνεργασία και με την Επιτροπή Γεωργίας έτσι ώστε να γίνει ε, αξιολόγηση για το κατά πόσον ε, θα είναι απαραίτητη μία αποστολή επιτόπου. Δεν λήφθησαν άλλες αποφάσεις στη διάρκεια της συνεδρίας των συντονιστών και επομένως το σημείο 16 ολοκληρώθηκε και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 17 της ημερησίας διατάξεως είναι η αναφορά 0874 του 2013 που έχει υποβληθεί από την Ροζέλα Τζάτσι ε, με άλλες 33 συγγνώμη, υπογραφές ε, σχετικά με την οργάνωση του τοπικού συστήματος υγείας, κυρίως δε σχετικά με το κλείσιμο ενός ε, νοσοκομείου στην περιφέρεια της Καλαβρίας στην Ιταλία ε, σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε τοπικό επίπεδο. Η υπογράφουσα είναι εδώ την συνοδεύει δε ο αντιδήμαρχος Ανδρέα Πέτα, καθώς επίσης και ο δόκτωρ Δομένικο Ταλαρίκο. Θα δώσω το λόγο στην υπογράφουσα, την κυρία Τσάτσι, έτσι ώστε ε, σε πέντε λεπτά να μας μιλήσει για την αναφορά αυτή. Παρατηρήσει εκτός μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς. Ναι, δεν ήξερα τι να κάνω κι εγώ. Ε, δεν ε, είχα καταλάβει ότι είσαστε εδώ. Ναι, είναι παρόν και ο δήμαρχος του Τρεμπιζάτσε. Το λόγο έχει η κυρία Ροσέλα Τσάτσι. Ευχαριστώ πολύ σε όλους σας. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη ευκαιρία για μας και η δυνατότητα να παρουσιάσουμε ανοιχτά τη θέση μας με τις τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές και να πάρουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί. Λέγομαι Ρόζα Λατσάτσι και έχω αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία μαζί με τον Δήμαρχο και άλλους τοπικά εκλεγμένους που υπέγραψαν αυτή την αναφορά. Εκπροσωπούμε 3.000 πολίτες, εδώ παρόντες. Είναι ο αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Πέτα και ο κ. Σταλαρίκο, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και ο δήμαρχος του Τρεμπιζάτσε. Έχουμε κάποια μια παρουσίαση PowerPoint για να σας παρουσιάσουμε την κατάσταση και τώρα θα μιλήσω τελικά. Η περίπτωση αυτή εντάσσεται σε μια καταστροφική υγειονομική κατάσταση που ε, ε, βλέπει στην περιφέρεια της Καλαβρίας να γίνονται τρομερές περικοπές όσον αφορά την υγεία. Ε, υπάρχει ένα, μια τρύπα στον προϋπολογισμό 1,5 δις ευρώ και σήμερα κλείνουν μέσα στο Τρεμπισάτσε διάφορες υγειονομικές δομές οι οποίες άρχισαν να κλείνουν από το 1985 και μετά. Ah, οι υγειονομικέ δομέ ε, λοιπόν ε, ε, καλή ποιότητα, οι οποίε, αφού δημιουργήθηκαν εγκατελείφθησαν το Ιταλικό κράτος έχει δαπανίσει 14 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια. Εν τω μεταξύ όμως είναι πολλοί οι πολίτες ε, οι οποίοι ε, για να θεραπευθούν θα πρέπει να πάνε μακριά. Η περίπτωση αυτή του νοσοκομείου του Τρεμπιζάτσε ε, μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ε, διότι ε, μιλάμε για μια περιοχή με 17 ε, δήμους και περισσότερες από 5.000 τουρίστες το καλοκαίρι. Σε πολλές περιπτώσεις όμως έχουμε πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα όσον αφορά το οδικό δίκτυο και βλέπετε εδώ και το δικό δίκτυο της περιοχής. Μια μισή ώρα χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στο πρώτο σημείο, στο βοηθειών. Ε, ε, ε, ένας αγώνας εναντίον του χρόνου στην ουσία γιατί η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και τη στιγμή που θα αναλάβει, θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή ξεκινάει μια άλλη αναζήτηση μάταια για κλίνη ελεύθερη σε κάποια από τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Και από οικονομική καθαρά άποψη αυτή, αυτό το κλείσιμο του νοσοκομείου του κοστίζει περισσότερο παρά ε, οδηγεί σε κάποια αποταμίευση. Ε, το κόστος ε, της κινητικότητας από τα 2 εκατομμύρια ευρώ το 2009 πέρασε στα 9 εκατομμύρια ευρώ το 2010 για την ε, ε, περιφέρεια, ε, κυρίως δεν λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές φορές πρέπει να πάμε στη γειτονική περιφέρεια της Μπαζιλικάτα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσαμε, μια και δεν μπορέσαμε σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο να βρούμε το δίκαιο μας, να περάσουμε στην επόμενη ταχύτητα που είναι βεβαίως το ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αναφορά στην Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, ε, που αναφέρεται στην υποχρέωση, συγκεκριμένα στο άρθρο 4, η υποχρέωση για την παροχή υγείας. Αναφέρεται λοιπόν ότι κάθε, κάθε πολίτης έχει δικαίωμα σε πρόσβαση στην περίθαλψη καθώς επίσης και σε μια υγειονομική περίθαλψη η οποία θα είναι καλού επίπεδου. Επίσης το άρθρο 168 της συνθήκης Ευρωπαϊκής λειτουργίας αναφέρεται ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, έχει την υποχρέωση να συνδυάζει τις πολιτικές και να ολοκληρώνει τις εθνικές πολιτικές καθώς επίσης και να αποβλέπει στην βελτίωση της δημόσιας υγείας. Είναι επομένως σαφές ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επικουρικός. Στην ουσία δηλαδή δεν παρεμβαίνει όσον αφορά την οργάνωση ε, των υπηρεσιών υγείας ε, αλλά ε, θα πρέπει να στηρίξει μέσω παρεμβάσεών της περιπτώσεις σημαντικής έλλειψης σε αυτήν την ε, περίπτωση ε, η αναφορά λοιπόν αναλαμβάνει έναν ρόλο καταγγελτικό όσον αφορά τη διαχείριση της ε, υγείας η οποία δεν σέβεται την αρχή που μόλις ανέφερα. Όσον αφορά την αρχή αυτή και έτσι ώστε η χώρα να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έχει την τάση να αποκεντρώνει τη διαχείριση ε, σε μια οπτική ενδεχόμενης βελτίωσης της οικονομικής ε, κατάστασης. Αλλά ε, σε μερικές περιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες και οι εξειδικεύσεις της κοινότητας αναφοράς. Αυτό ίσχυσε και στη δική μας περίπτωση όπου έχουν απογυμνοθεί όλες οι υπηρεσίες υγείας ακόμα και οι υπηρεσίες σε πρωτοβάθμιο ε, επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην υγεία που σημαίνει ότι προσφέρονται, παρέχονται οι απαραίτητες δραστηριότητες και υπηρεσίες. Ε, αυτές ε, οι υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να είναι ίδιες για όλους. Και βεβαίως δεν αναφέρουμε μονάχα στους Ιταλούς πολίτες, στους ντόπιου, αλλά και στους τουρίστες, Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μας το καλοκαίρι καλοκαίρι. Επίσης θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, και την ανάγκη όλοι όσοι ε, ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να έχουν το ίδιο ε, επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο είπαμε ότι θα πρέπει η ενωσιακή νομοθεσία να μεταφέρεται με τρόπον ώστε να παρέχονται σωστά οι υπηρεσίες υγείας και έτσι ώστε να μην ενθαρρύνονται οι πολίτες να αναζητούν υπηρεσίες υγείας καταλληλότερες πέραν των συνόρων σε αυτή την περίπτωση όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή οι πολίτες της ε, περιοχής αυτής υποχρεώνονται ή ενθαρρύνονται ε, να αναζητήσουν υπηρεσίες υγείας εκτός των συνόρων. Ε, νομίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν η ενθαρρυνονται να αναζητησουν υπηρεσιες υγειας εκτος των συνορων νομιζουμε οτι δεν ειναι δυνατον η ευρωπη να μην ακούσει προσεκτικά το αίτημά μας. Ε, δεν είναι δυνατόν να παραμείνει απαθής σε αυτήν την καταγγελία ε, των ε, πολιτών της περιοχής μας. Δεν είναι δυνατόν ε, να παραμείνει η Ευρώπη μακρινή στον πολίτη. Θα πρέπει να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στην περιοχή αυτή απαιτούν το δικαίωμα να υπάρχουν κρεβάτια για επίγουσες περιπτώσεις. Και αυτό έχει επιπτώσεις στην πολιτική για την υγεία στην Καλάμπρια. Χρειάζεται διαφάνεια για τη χρήση των ενωσιακών πόρων. Σε τελευταία ανάλυση εγγυώνται στην πράξη, είναι εγγυημένα στην πράξη τα δικαιώματα των πολιτών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία. Ευχαριστώ κυρία Τσάτσι. Ο κύριος Γκέραλτ Χέγκεντορφ ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Να σας παρουσιάσω την άποψη της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Δηλαδή, ποιος είναι αρμόδιος για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Αναφερθήκατε στο άρθρο 168 που αφορά τις πολιτικές υγείας. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι συνδέεται ιδιαίτερος με την ιατρική περίθαλψη και την κατανομή πόρων που επίσης ε, στον ένα τον άλλο βαθμό σχετίζεται με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού και εδώ θεωρούμε ότι αναφέρεται σαφώς ότι οι τομείς αυτή πολιτικής είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και η λήψη μέτρων για τους τομείς αυτούς και η χρηματοδότησή τους. Αναφερθήκατε επίσης στο άρθρο 35 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που εστιάζει στην αρχή ότι όλα τα μέτρα προληπτικής υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών στην ε, ιατρική περίθαλψη υψηλού επίπεδου βασίζονται σε εθνικές αρχές και πρακτικές. Και εδώ λοιπόν ε, πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Πυρίλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Ροσέλα Τσάτσι, η οποία μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσουμε για ένα πρόβλημα ε, το οποίο, όπως μας περιέγραψε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν εμπίπτει στις θερμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αναμφίβολα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ε, για την ε, ε, υγεία στην Καλαβρία. Καταλαβαίνετε ότι όταν μια τόσο σημαντική δομή κλείνει, αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Έχουμε εδώ έγκριτους εκπροσώπους της περιφέρειας αλλά και της πόλης του Στρεμπιζάτσε και είμαστε όλοι εδώ για να στηρίξουμε με μεγάλη ρόμη αυτή την αναφορά. Αγαπητή θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και την πρόεδρο ε, η οποία απεφάσισε ότι ακόμα και με την αρνητική ε, ε, απόφαση της Επιτροπής αποφάσισε να συζητήσουμε παρόλα αυτά για ένα πρόβλημα το οποίο ίσως είναι πρόβλημα της Καλαβρίας. Η πρόεδρος έρχεται και αυτή από περιφέρεια του Νότου, από τη μεσημβρινή Ιταλία και γνωρίζει τα προβλήματα ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσει το κράτος μέλος και προκειμένου η περιφέρεια της ε, ε, Καλαβρίας μαζί με τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο ε, ξέρω ότι θα συνεχίσετε τις προσπάθειες και αν και η πρόεδρος Ματσόνη έκανε μια κίνηση ε, στη, ε, προς την περιφέρεια της Καλαβρίας δεν θα έκανε κακό. και από την άλλη πλευρά είναι πολύ σημαντικό που η Ρωσέλα μάζεψε τόσες υπογραφές για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο προσφυλές σε όλους τους κατοίκους της περιοχής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Ακούσαμε τον αναφέροντα και την Κομισιόν και είναι πάντοτε το θέμα ποιος έχει αρμοδιότητα. Αυτό που μας λείπει βεβαίως στην όλη ιστορία είναι η τοποθέτηση και η περιγραφή της κατάστασης θα μπορούσαμε ίσως να πούμε και την υπερασπιστική γραμμή της ίδιας της περιφέρειας ή της ε, εθνικής κυβέρνησης που είναι υπεύθυνη. Οπότε θα ζητούσα από την Κομισιόν να, το πω έτσι, η περιφερειακή κυβέρνηση ε, να, ζητήσει η Κομισιόν από την περιφερειακή κυβέρνηση ε, μια περιγραφή της κατάστασης από ό,τι λένε οι αναφέροντες δεν εξασφαλίζεται πλέον η προεπληκτική υγεία, η Κομισιόν λέει ότι δεν είναι αρμόδια, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα γεγονότα. Οπότε πρέπει να μάθουμε από την ίδια την περιφέρεια τι συμβαίνει και γι' αυτόν τον λόγο να κρατηθεί ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Γιάρ. Δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο, δράτω όμως της ευκαιρίας για να επαναλάβω μία αρχή η οποία επανειλημμένα έχει αναφερθεί στις εργασίες της Επιτροπής μας. Έχουμε μία διαδικασία έτσι ώστε ε, να γίνει παραδεκτή μία αναφορά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες οι οποίοι βεβαίως έχουν ε, και ένα ευρύ περιθώριο ερμηνείας. Ε, ε, γιατί η Επιτροπή είναι εδώ για να ακούει τα προβλήματα των πολιτών που αφορούν όλα τα πεδία της της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Εδώ αναφερόμαστε σε μία αρχή η οποία ρητά αναφέρεται στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας η Επιτροπή ε, αναφορών ε, ασχολήθηκε πολλές φορές ε, με θέματα τα οποία ε, θεωρούν τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων σε, συνδυασμό μάλλον και με την συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν βασική νομοθεσία και επομένως άνοιξε ένα πεδίο πιο ευρύ όσον αφορά τις δραστηριότητες της εν λόγω Επιτροπής. Τέλος, υπάρχει και μια στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία διαπιστώνουμε σε πολλές περιπτώσεις ε, η οποία κατά την άποψή μας και το έχουμε πει επανειλημμένα απορρίπτει την πλήρη εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας ε, ε, και αυτό αμφίδρομα γιατί η αρχή της επικουρικότητας λέει ότι θα πρέπει να δοθεί στο, θεσμικό επίπεδο το πιο κοντινό στον πολίτη η απάντηση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε περίπτωση που δεν καλύπτεται αυτό από το τοπικό επίπεδο θα πρέπει κανείς να ανεβεί την θεσμική κλίμακα μέχρι ότου φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να δώσει απάντηση στον προβληματισμό των πολιτών. Επομένως δεν είναι δυνατόν εμείς να αφήσουμε ακάλυπτα τα δικαιώματα των πολιτών, ιδιαιτέρως δε τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Πιστεύω ότι είναι σωστό να δεχτούμε την πρόταση που ακούστηκε, να ε, στείλουμε επιστολή λοιπόν όπως έχουμε επανειλημμένα κάνει στην περιφέρεια της Καλαβρίας ζητώντας αναφορά της καταγγελθήσης καταστάσεως. Και επίσης να στείλουμε επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό της Εθνικής Κυβερνήσεως έτσι ώστε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση. Ε, γιατί ξεκινούμε από ένα και μόνο σημείο εκκίνησης που είναι ε, ε, η υποχρέωση προστασίας των πολιτών από πλευρά των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Η κυρία Τσάτσι. Δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι μετά από την ε, συζήτηση που έλαβε χώρα ε, η Επιτροπή εδώ δέχτηκε ε, την αναφορά μας βασιζόμενη σε μία ε, πραγματική ευρωπαϊκή στάση. Στάση η οποία ε, πρέπει να είναι υπεύθυνη απέναντι σε ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο όμως παραμερίζεται ε, τώρα. Ε, θεωρούσαμε ότι θα έκλεινε αυτή η αναφορά ε, και τώρα αναπτερώνεται το ηθικό μας ε, και η ελπίδα μας ότι θα μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και ταυτόχρονα αναπτερώνονται και οι ελπίδες μας όσον αφορά την καλή αντιμετώπιση των πολιτών από πλευράς των θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι αυτό είναι καλό και για μας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την αναφέρουσα, τους υπογράφοντες, τους παρισταμένους. Ε, και βεβαίως θα κάνουμε όπως είπαμε προηγουμένως θα στείλουμε επιστολή στις αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές αρχές ε, όπου θα αναφέρουν, θα ζητούμε διευκρινήσεις σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν κάνει οι πολίτες. Βεβαίως μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές θα προχωρήσει το θέμα. Πάρα πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως είναι η αναφορά υπαριθμών που έχει εγγραφεί μάλλον στο ε, σημείο 18 της Μερισίας Διατάξεως. Είναι η αναφορά 0319 του 2013 από τον Αλεσάνδρο Τσαμπρόνε ε, και εξ ονόματος του δικτύου ενώσεων του Καστέλ Βολτούρνο σχετικά ε, με περιβαλλοντικές ζημίες στην περιοχή της προαναφερθήσας κοινότητας ο αναφέρον δεν είναι παρόν. Ε, έχει στείλει όμως στην Προεδρία λεπτομερές έγγραφο σχετικά με την αναφορά του, σχετικά με τις ε, καταγγελίες του, ε, καθώς επίσης και επικαιροποιημένα στοιχεία για την λόγο καταγγελία, τα οποία έχουν διανεμηθεί. Θα δώσω άμεσα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ζιλ Ντελάγιο. Ευχαριστώ. τα περιβαλλοντικά εγκλήματα ανησυχούν ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της καταπολέμησης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα θεωρούνται ως ε, αναδιόμενη απειλή στα πλαίσια της Ένωσης στα πλαίσια αυτού που αποκαλούμε πολιτικό κύκλο για την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματο, του οποίου νέε προτεραιότητε για την περίοδο 14-17 μόλι καθορίστηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει λοιπόν να χρηματοδοτήσει προγράμματα για το θέμα αυτό. Αυτά γενικά. Τώρα για την ε, συγκεκριμένη αναφορά και τα θέματα που θέτει. Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει ε, να σέβονται την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα οργανωμένα και συγκεκριμένα τα περιβαλλοντικά εγκλήματα το οποίο περιβάλλει τον ορισμό των ποινών και των αδικημάτων για τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα την απόφαση πλαίσιο του 2008 για το οργανωμένο έγκλημα και την οδηγία του 2008 για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω ποινικού δικαίου. Αυτά είναι τα εισαγωγικά σχόλια που θέλουμε να κάνουμε από αυτού του θέματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έδωσε ένα γενικό πλαίσιο, χωρίς όμως να μας βοηθήσει έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε ε, στα ερωτήματα των πολιτών που απευθύνθηκαν σε εμά. Ο συνάδελφος Γιάρ ήθελε όχι, δεν θέλει το λόγο. Α, ναι, εντάξει. Δύο πράγματα. Ο αναφέρον ε, παραπονείται για ε, αποζημίωση στην περιοχή και ταυτόχρονα εγώ θα ήθελα να μάθω ποια είναι η κατάσταση ε, θυμώνω λίγο όταν ακούμε απαντήσεις από την Κομισιόν χωρίς να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να διαπιστώσουμε ποια, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία. Δεν μπορώ να αξιολογήσω εγώ από εδώ. Υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, ή δεν υπάρχουν. Έχουν γίνει κάποιες μετρήσεις από δημόσιες αρχές. Συνήθως οι δημόσιες αρχές ε, υποχρεούνται να ε, διαπιστώνουν ποια είναι η κατάσταση ή περιβαλλοντική. Δεύτερο μέρος, ε, στο δεύτερο μέρος η Κομισιόν προσπάθησε να απαντήσει. Λέει εδώ ότι αυτές οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενισχύονται από το εργανωμένο έγκλημα και την παράνομη μετανάσταση. Θεωρώ δεδομένο ότι όταν, τα δημόσια, όταν οι δημόσιε αρχέ διαπιστώνουν περιβαλλοντική υποβάθμιση θα πρέπει να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα. Οπότε μου φαίνεται κάπω σύντομη, ανεπαρκή ε, και για μένα προσωπικά κάπω μη ικανοποιητική η απάντηση τη Κομισιόν. Ποιο είναι το συμπέρασμα, Τα πράγματα λοιπόν είναι καλά. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι ο αναφέρον δεν θα υπέβαλε αυτή την αναφορά αν τα πράγματα ήταν καλά. Οπότε νομίζω ότι Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι δεν πολύ καταλαβαίνω και δεν με ικανοποιεί η απάντηση της ε, Κομισιόν. Ε, Θα μπορούσα μάλιστα να προσθέσω ότι προκύπτει από την ε, συγκεκριμένη αναφορά ότι σε αυτήν την συγκεκριμένη περιφέρεια υπάρχει η λεγόμενη μεγαλύτερη χωματερή ε, της ε, Ευρώπης. Ε, αν προσθέσουμε σε αυτό τα όσα καταγγέλει ο αναφέρον σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, σχετικά με την πλήρη εγκατάλειψη της περιοχής όσον αφορά, την, όσον αφορά τα απόβλητα, πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καταδικασμένη αδίκωση η Ιταλία για τέτοιες περιπτώσεις και εν πάση περιπτώσει λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά θα περιμέναμε μια διαφορετική αντίδραση της <clears throat> Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, αναφερόμενοι σε αυτά που μόλις μας είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερωτώ, υπάρχουν ε, δυνατότητες και πόροι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη πληγή του οργανωμένου εγκλήματος ε, κυρίως όσον αφορά περιβαλλοντικά εγκλήματα ε, γιατί η Ιταλία ξέρουμε ότι ζήτησε και έλαβε ενωσιακούς πόρους ε, για το θέμα αυτό. Υπάρχουν επίσης πόροι για την εξυγίανση και αποκατάσταση των χώρων που παλιότερα ήταν χώροι υγειονομικής ταφής ή χωματερές ε, και οι οποίες όμως δεν κάλυπταν τις συμβατικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα όσον αφορά την αποκατάσταση και εξυγίανση. Όλοι οι πολίτες και οι συγκεκριμένοι πολίτες της περιοχής έχουν δικαίωμα ε, για προστασία της υγείας τους. Αλλά δεν κυδεμονεύεται αυτή η προστασία στην προκείμενη περίπτωση. Και έστω και αν ε, εν προκειμένου η αρμοδιότητα είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των κρατών μελών θα έπρεπε να υπάρχει πιο συγκεκριμένος και πιο ε, σαφής ρόλος ελέγχου από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό που σας λέω τώρα θέλετε να μου απαντήσετε. Äh, Ήθελα να πω ότι αν έχουν δοθεί ε, ευρωπαϊκοί πόροι, ενδεχομένως αυτές οι προφορές θα έπρεπε να διατεθούν και στην ε, Επιτροπή του Προϋπολογισμού. Ε, να γίνει δηλαδή ένας έλεγχος αφού δόθηκαν χρήματα ευρωπαϊκά, αν τελικά έφτασαν στον προορισμό τους και αν χρησιμοποιήθηκαν με τον τρόπο ε, για τον οποίο προορίζονταν. Και ε, ε, αν έχουν δοθεί ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα πράγματα και η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα με ενδιέφερε λοιπόν κάτι τέτοιο. Grazie. Mr. Σας ευχαριστώ, κύριε Τερπελάγιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για τα συγκεκριμένα προγράμματα για να καταπολεμηθεί το περιβαλλοντικό έγκλημα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπό τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές η Κομισιόν προτίθεται να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα προγράμματα είναι ένας νέος τομέας θεματικής πολιτικής της Ένωσης και επίσης ε, και το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια θα χρηματοδοτήσει την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προ, προ, εγκλημάτων. Για το δεύτερο θέμα, για τα εσωτερικά, από τον τομέα εσωτερικών υποθέσεων τα κράτη-μέλη με βάση την ενωσιακή νομοθεσία έχουν την υποχρέωση να αντιμετωπίσουν το σοβαρό περιβαλλοντικό έγκλημα με αποτελεσματικά ανάλογα με το πρόβλημα μέτρα. Αλλά αυτή η νομοθεσία δεν δημιουργεί υποχρεώσεις για την εφαρμογή κυρώσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι περιορισμένο λοιπόν το κοινοτικό κεκτημένο σε αυτό το τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει με μονομένες περιπτώσεις όπως αυτή. Ωραία. Ευχαριστώ παρόλα αυτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έστω και αν οι απαντήσεις παραμένουν ασαφείς και γενικόλογες σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα. Θα πρέπει και πρόκειται να μείνει ανοιχτή η αναφορά ε, ενώ θα ζητήσουμε όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ζητήσει με πιο συγκεκριμένο τρόπο σχετικά με τους, ε, τις συγκεκριμένες ε, περιοχές, δηλαδή να μας δώσει γραπτή απάντηση την οποία δεν έχουμε λάβει μέχρι τώρα, αλλά θα ζητήσουμε και από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ε, να ε, κάνει μια επαλήθευση όπως ζήτησε και άλλος το συνάδελφος Γιάρ σχετικά με τους ευρωπαϊκούς πόρους, τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία ενδεχομένως δόθηκαν ε, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος έτσι ώστε να προχωρήσουν διαδικασίες οι οποίες συνδέονται με την αναφορά. Κυρίως δεν να μάθουμε πώς, με ποιο τρόπο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια αυτά γιατί η κατάσταση μας αφήνει να να ε, υποψιαστούμε, να υποπτευθούμε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ίσως τα ή ίσως και καθόλου τα ε, ε, κονδύλια αυτά το οφείλουμε αυτό στους πολίτες οι οποίοι απευθύνονται σε εμά έτσι ώστε να προστατέψουν τα δικαιώματά τους. Περνάμε στην επόμενη αναφορά, είναι η 304 του 2013, αναφορά του κυρίου Λορέντσο Φοντάνα ο οποίος θα έπρεπε να είναι παρόν. Α, εδώ είστε. Δεν σας είδα. Κρυφτήκατε. Δεν σας είδα, ζητώ συγγνώμη. Είναι παρόν λοιπόν ο συνάδελφος Λορέντζο Φοντάνα. Του δίνω το λόγο για πέντε λεπτά έτσι ώστε να ε, αναφερθεί στην συγκεκριμένη αναφορά. Δεν είμαι και μικροκαμωμένος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η αναφορά που υπέβαλα μαζί με πολλούς συνυπογράφοντες αφορά ε, μια πολύ δύσκολη κατάσταση ε, του σοφρονιστικού συστήματος. Όπως ξέρετε είναι πολλές οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα κυρίως όσον αφορά τον συνοστισμό στις φυλακές. Ε, από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο υπερβολικός συνοστισμός στις φυλακές έχουμε και έκπτωση της, ε, ε, της αξιοπρέπειας των εγκλήστων. Γι' αυτό ακριβώς ε, ζητούσαμε, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, την δυνατότητα να υπάρξει μια στρατηγική βάση της οποίας ε, να επιστρέφουν στη χώρα καταγωγή τους οι καταδικαστέντες. Στα πλαίσια αυτής της πρότασης θεωρούμε ότι θα αντιμετωπιστεί καλύτερα το θέμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των ανθρωπίνων αυτών. Επίσης, εάν επιστρέψουν στους, στις χώρες καταγωγής τους τα πρόσωπα αυτά, ίσως να έχουν και μια καλύτερη ε, αντιμετώπιση. Και αυτό να αφορά και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τρίτες χώρες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ξεκίνησαν κάποιες τέτοιες διαδικασίες. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι εάν ε, υπάρξει ενωσιακή στρατηγική στον τομέα αυτό ε, θα έχει οπωσδήποτε μεγαλύτερο βάρος από ότι κάποια μέτρα που αναλαμβάνει μόνη της μια μεμονωμένη χώρα μέλος. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα του συνοστισμού στις φυλακές ε, είναι ένα κοινό πρόβλημα σε όλες τις χώρες μέλη και η καθεμία προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα του ε, συνοστισμού στις φυλακές με διατάξεις οι οποίες είναι πρόσκαιρες, λειτουργούν για μερικούς μήνες αλλά η κατάσταση δυστυχώς επιστρέφει στα αρχικά επίπεδα ε, πάρα πολύ ε, γρήγορα. Με αυτό το σκεπτικό υποβάλαμε τούτη την αναφορά. Ελπίζουμε δε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί παραδεκτή και να φτάσουμε σε κάποια ενωσιακή νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φοντάνα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον λόγο έχει η κυρία Τζέσικα Μπενέσερ. Um, Ευχαριστώ. Υπάρχει μια απόφαση πλαίσιο 909 για την ασφάλεια και, την εσωτερική, και τις εσωτερικές υποθέσεις του 2008 για την επιστροφή των φυλακισμένων σε κάποιο άλλο κράτος μέλος με το οποίο, στο οποίο διέμεναν ή το οποίο είναι κάτοικοι ή έχουν στενούς δεσμούς για να εκτίσουν εκεί τις ποινές με στόχο την κοινωνική τους αποκατάσταση. Η απόφαση αυτή προβλέπει δυνατότητα τέτοιων μεταφορών ακόμη και χωρίς τη συνένεση του εγκλήστου στην χώρα προέλευσής του στις εξής περιπτώσεις. Πρώτον, ο καταδικασμένος πρέπει να είναι πολίτης ε, του κράτους αυτού και να ε, διαμένει στο κράτος αυτό για να σταλεί χωρίς τη συνένεσή του. Δεύτερη δυνατότητα να σταλεί πίσω στη χώρα είναι, χωρίς συνένεση, είναι εάν ούτως ή άλλως επρόκειτο να απελαθεί προς τη χώρα αυτή μετά τη λήξη της ποινή του. Και η τρίτη δυνατότητα για ακούσια επιστροφή είναι αν έχει ήδη δραπετεύσει στη χώρα του. Αυτά λέει το άρθρο 6 της απόφασης πλαίσιο. Ωστόσο η απόφαση πλαίσιο αυτή δεν έχει εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη παρά το ότι η προθεσμία για την ε, εφαρμογή της έληξε την 5η 12 του 2011. Ήδη μέχρι στιγμής 18 κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει αυτή την απόφαση πλαίσιο. Η Επιτροπή ενέκρινε μια έκθεση για την εφαρμογή αυτής της απόφασης πλαίσιο στις 5 Δευτέρου τρέχοντος. Εφόσον και τα δύο κράτη-μέλη τα οποία θα μπορούσαν να εμπλακούν σε τέτοια μεταφορά δεν έχουν εφαρμόσει αυτή την οδηγία, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομικό καθεστώς όπως η Σύμβαση του 1988 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μεταφορά των ε, φυλακισμένων και το συμπληρωματικό πρωτοκόλλο του 1997 με το συμπληρωματικό πρωτόκολλο μια τέτοια μεταφορά μπορεί να γίνει χωρίς τη συνένεση του ε, καταδίκου. Αυτό το συμπληρωματικό πρωτόκολλο επικυρώθηκε από 26 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων και των περισσότερων κρατών της Ένωσης. Αυτές οι διαδικασίες ρυθμίζονται μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που ε, έχουν συνάψει τα κράτη-μέλη ή μέσω της προαναφερθήσης συμβάσεω του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου. Η σύμβαση αυτή είναι του 1983. Ε, έχει επικυρωθεί από 63 κράτη-μέλη. Καταλήγοντας, και η απόφαση 2008 κάθε 909 και το συμπληρωματικό πρωτόκολλο του 1997 στην Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 1983 ήδη αποτελούν ένα πλαίσιο που μπορούν να επιτρέψουν την έκθεση ποινών στη χώρα προέλευσης των καταδικαστέντων με βάση μια δικαστική απόφαση μπορεί και ακουσίως να μεταφερθούν. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνεται και αυτομάτως. Διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παράγων κοινωνικής αποκατάστασης και επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ε, αμφισβητήσουν αν δεν συμφωνούν με την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Ο συνάδελφο Φοντάνα. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ωστόσο, κατά την άποψή μου εδώ, το πρόβλημα έγκυται στο ότι συχνά πρόκειται για διμερείς ε, συμφωνίες, ε, οι οποίες δυστυχώς ε, ποικίλουν από χώρα σε χώρα, διαφέρουν από χώρα σε χώρα είναι καλό να υπάρχουν αυτές ε, οι διμερείς ε, ε, συμφωνίες και είναι σαφές. Από την άλλη πλευρά εξίσου σαφές είναι ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει αυτόν τον ενωτικό της ρόλο σε, και όσον αφορά τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και όσον αφορά τρίτες χώρες με τις οποίες δεν έχει τέτοιες συμφωνίες. Εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας κανονισμός ε, ο οποίος να ισχύσει για όλες τις χώρες. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή εν αναμονή ε, γραπτής απάντησης της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, έτσι ώστε να δούμε ακριβώς ε, πώς θα έχει ο κανονισμός αυτός γιατί πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να πιέσουμε τις χώρες μέλη οι οποίες ακόμα δεν έχουν υπογράψει την απόφαση πλαίσιο και που ακόμα βρίσκονται σε ε, ε, ελλειπή διαδικασία όσον αφορά αυτό το θέμα. Πίτερ Εκτός μικροφώνου. Αν κατάλαβα καλά, ο αναφέρον ζητά να υπάρχει ένας κανονισμός ή ε, θεωρεί τέλος πάντων ότι η απόφαση πλαίσιο αυτή δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Ο αναφέρον επίσης ανέφερε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ε, διμερείς συμφωνίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο θα ε, ε, ζητούσα ναι, γνωμοδότηση Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για το αν θεωρεί ότι υπάρχει όντως μια τέτοια κατάσταση. Ως ε, Ευρωκοινοβούλιο έχουμε αυτό το έμεσο δικαίωμα υποβολής αιτήματος. Αν το Κοινοβούλιο λοιπόν Θεωρήσε ότι εδώ απαιτείται κάποια νομική πράξη, τότε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα έμεσης υποβολής ε, αιτήματο στην αρμόδια. Δεν είμαι νομομαθής ε, εγώ προσωπικά, είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο ή όχι ή ε, θα αρκούσε η εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο. Τίθεται και βέβαια και το ερώτημα για ποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση πλαίσιο και είπε ο αναφέρον ότι τουλάχιστον για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, να περιλαμβάνονται όλες αυτές οι προβλέψεις σε κανονισμό. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω, αλλά θα μπορούσαμε τέλος πάντων να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό και με τον τρόπο που ανέφερε. Πρόεδρος, προσθέτω ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έστειλε ε, έκανε μια αποστολή την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία ακριβώς για να ασχοληθεί και να επιβεβαιώσει τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην αναφορά και θα συζητηθούν περαιτέρω τη 10η Απριλίου. Η έκβαση λοιπόν της αποστολής ε, ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και εν αναμονή και των συμπερασμάτων της εν λόγω αποστολής θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα στοιχεία από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, θα πρέπει να έχουμε την γραπτή απάντηση με τα συγκεκριμένα ε, στοιχεία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διαπιστώσουμε εάν και η Ιταλία αλλά και άλλες ε, χώρες ε, δεν ε, έχουν δείξει την απαιτούμενη πειθαρχία όσον αφορά την την εφαρμογή του κανονισμού και τη μεταφορά του κανονισμού αυτού, την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και για την Ιταλία λέω αλλά και για άλλες περιπτώσεις χωρών ε, γιατί ξέρουμε ότι επανειλημμένα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποστείλει μομφές προς την ε, ε, Ιταλία και την Ιταλική κυβέρνηση για, τα, για παρόμοια θέματα. Αλλά βεβαίως εδώ δεν μπορούμε να απαντήσουμε στους αναφέροντες απλώς λέγοντας ότι έχει επικριθεί η χώρα επανειλημμένα για τα θέματα αυτά. Οι αναφέροντες και οι υπογράφοντες στην αναφορά χρειάζονται πιο συγκεκριμένα συγκεκριμένη απάντηση, απάντηση με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Φοντάνα για την αναφορά που έχει υποβάλει, γιατί όταν έχουμε συναδέλφους οι οποίοι υποβάλλουν αναφορές, τότε ε, δυναμώνει οπωσδήποτε και ο ρόλος, ο θεσμικός ρόλος της Επιτροπής Αναφορών. Ευχαριστώ λοιπόν και τον συνάδελφο, αλλά και όλους τους πολίτες που έχουν υπογράψει την αναφορά αυτή. Ολοκληρώνεται το θέμα αυτό. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξης πράξεως είναι η αναφορά 357 του 2012, ε, αναφορά του κυρίου Γιάνν Φλωρί, ε, Γάλλου υπηκόου, ο οποίος δεν είναι παρόν, αλλά θα εκπροσωπηθεί από την συνάδελφο κυρία Μπελιέ, ε, στην οποία δίνω και το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι αναφέροντες δεν μπορούν να είναι παρόντες σας παρακαλούν να τους συγχωρήσετε και με παρακάλεσαν να διαβάσω το εξής μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα του Γιάνν Φλωρή και του συνόλου των αναφερόντων που απευθύνθηκαν στην Επιτροπή μας. Κάτω τον Απρίλιο του 2014 ο κύριος Ντόρισον που είναι υπεύθυνο ε, ε, για ε, την επιχείρηση στο Καμίν θα στείλει στον Υπουργό Οικολογίας και Ανάκαψης της Παραγωγής την έκθεσή του και θα κάνει προτάσεις για να εξηγήσει την απόφασή του. Η διαβούλευση έγινε μεταξύ της 15 του 2013 και της 15 Φεβρουαρίου 2014. Υποβλήθηκαν 26 ε, αιτήματα, 26 ε, προτάσεις, από τα οποία 23 είναι κατά αυτής της προσπάθειας. Καθ' όλη τη διαδικασία διαβούλευσης ο υπεύθυνο για την εκαθάριση, κ. Ντελέ, θεωρεί ότι ο καλύτερος, η καλύτερη λύση θα ήταν να περιοριστούν οι ουσίες αυτές και παρά το ότι υπάρχει κίνδυνος ε, μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα λέγεται ότι ποτέ δεν θα είναι μη πόσιμο το νερό αλλά πώς μπορούμε να ξέρουμε ποιο θα είναι το όριο ποσιμότητα σε 100 ή 300 χρόνια Εάν ε, απομακρύνουμε εντελώς τα απορρίμματα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εγγυηθούμε την ποσιμότητα του ύδατος και τον υδροφόρο ορίζοντα. Όλοι γνωρίζουν ότι τα φράγματα μπεντονίτη στην ουσία απλώς θα επιβραδύνουν την αναπόφευκτη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να απευθυνθούμε για άλλη μια φορά στην Επιτροπή σας για να επιθυμίσετε στη γαλλική κυβέρνηση ότι εάν αποσύρει μόνο μία μόνο ένα τμήμα από τα ιδιαίτερα τοξικά χημικά απόβλητα, απόβλητα που βρίσκονται εκεί θα παραβεί τις οδηγίες για το είδωρ που έχουν στόχο να διατηρήσουν ε, τον υδροφόρο ορίζοντα και να επιτρέψουν να υπάρχει επαρκές ε, είδωρ για όλες τις χρήσεις και να είναι βιώσιμη η χρήση του με βάση την μακροχρόνια προστασία των υδατίνων πόρων. Γι' αυτό με βάση την αρχή της πρόληψης που αναφέρονται στο άρθρο 194 της συνθήκης η πολιτική της Ένωσης στο περιβάλλον έχει στόχο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Βασίζεται στην αρχή της πρόληψης και της προληπτικής δράσης. Στην αρχή της διόρθωσης, ε, στην πηγή όλων των προβλημάτων που μπορεί να προκύψει για το περιβάλλον και στην αρχή του ομολύνων πληρώνει. Πρέπει λοιπόν να επενθυμίσουμε στο γαλλικό κράτος ότι χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική απόφαση για το θέμα αυτό γιατί το διακύβευμα είναι το πόσιμο είδωρο του πληθυσμού της περιοχής και δεν πρόκειται απλώς για ένα ε, συνηθισμένο γεγονότος ε, ε, κλεισίματος ενός ορυχείου σε περίοδο κρίσης. Ευχαριστώ για την Κομισιόν τώρα ο κύριος Μπαλασάς Ούρμπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω και την ε, παλαιότερη θέση της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας αναφερθήκαμε στην οδηγία για τις χωματερές, για τους χώρους υγειονομικής ταφής, όπου υπάρχουν ε, κάποιες ε, απαιτήσεις που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υπεύθυνες αρχές, αλλά τελική απόφαση για την ε, δημιουργία και τη θέση και η εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, όλα αυτά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό αφορά και την οδηγία για τα υπόγεια ύδατα και για τα ύδατα που τονίζει ότι πρέπει να αποφεύγεται η επιδείνωση του υδροφόρου ορίζοντα και επίσης να είναι σε καλό επίπεδο μέχρι το 2015 τα ύδατα αυτά οι γαλλικές αρχές μετέγραψαν τις οδηγίες αυτές και έχουν και προγράμματα για τη διαχείριση των, ποταμίων λεκανών και επίσης έκαναν αναλυτική δημόσια διαβούλευση. Με βάση την πληροφόρηση που χορηγήθηκε στην Κομισιόν, οι γαλλικές αρχές γνωρίζουν τα προβλήματα και έχουν προτείνει και θα εφαρμόσουν μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι της οδηγίας και για να βελτιωθεί η κατάσταση. Τα μέτρα θα αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους. Δεν είναι θέμα απόφασης της Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν έχει δυστυχία που να καταδεικνύουν ότι τα μέτρα που προτείνουν οι γαλλικές αρχές θα έθεταν εν κινδύνο την εφαρμογή των στόχων της οδηγίας που προανέφερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο για το θέμα αυτό. Η κυρία Βελά. Δεν κατάλαβα πως άλλαξε η Προεδρία. Γι' αυτό με βλέπετε έκπληκτη. Σημείωνα και δεν είχα σηκώσει το κεφάλι. Ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσατε το λόγο. Αφού σας διάβασα το μήνυμα των αναφερόντων, να σας πω πώς το βλέπω εγώ το θέμα ως εκλεγμένη της περιοχής αυτής που έχει να κάνει με αυτό το χώρο ε, απόθεσης αποβλήτων στο Καμίν. Από το μήνυμα των αναφερόντων νομίζω ότι καταλάβατε την απογοήτευσή τους, την απόγνωσή τους. Είναι πολίτες, είναι ενώσεις που εδώ και χρόνια για το θέμα αυτό το έχουμε εδώ και δέκα χρόνια έχουν την εντύπωση ότι δεν ακούγεται η φωνή τους. Εκφράζουν δυσπιστία λοιπόν έναντι του ε, διευθυντή αυτής της επιχείρησης το Καμίν που δεν επιτρέπει ουσιώδη διάλογο για να ληφθεί σωστή απόφαση. Το γαλλικό κράτος χρειάστηκε 10 χρόνια για να αποφασίσει να παρέμβει και σήμερα μας παρουσιάζει μια λύση που θεωρούμε ανεπαρκή. Θεωρείται λοιπόν ανεπαρκής από τους περισσότερους στενά εμπλεκομένους εκτός, εκτός ίσως από την επιχείρηση την ίδια. Υπάρχει μια κινητοποίηση. Κατά τη διαβούλευση σε όλες τις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Στην τελευταία συνάντηση συμμετείχαν 200 άτομα. Υπήρξε διαβούλευση. Το τονίζει ο αναφέρον. Αλλά κατά τη διαβούλευση αυτή Και αυτό, όπως είπαμε, το λένε και 23 από τι 27 προτάσεις, οι αναφέροντες, οι ενώσεις τους, οι πολίτες, είχαν την εντύπωση ότι ευρίσκονται πρώτε Και αυτό τεκμηριώνεται από το ότι προτάθηκαν διάφορες λύσεις, αλλά η λύση της πλήρους ε, ε, απομάκρυνσης δεν περιλαμβανόταν. Και αυτό κυρίως καταγγέλει ο πληθυσμός, τα συνδικάτα το ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί η λύση της πλήρους απομάκρυνσης δεν λήφθηκε υπόψη. Παρά το ότι οι διάφοροι εμπειρογνώμονες και ιδιαίτερα ένας πολύ γνωστός εμπειρογνώμονας ο κύριος Μπεζέρ τονίζει ότι είναι δυνατό και ακόμη και αυτοί που προτείνουν την μερική απομάκρυνση αναγνωρίζουν ότι μπορεί ε, μακροπρόθεσμα να υπάρξουν επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ γιατί όπως θα θυμάστε τον Ιανουάριο 2013 ε, είχαμε ε, ακούσει τους ε, ενδιαφερομένους. Σας ευχαριστώ λοιπόν που το συζητάμε και τώρα. Είμαι πεπισμένη ότι η ακρόαση που έχουμε κάνει και η επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή μας έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να υπάρξει αυτή η διαβούλευση αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Εάν λοιπόν οι αναφέροντες επαυθύνονται και πάλι σε εμά και θέλουν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, είναι γιατί σε λίγο θα έχουμε τα πορίσματα αυτής της δημόσιας ε, διαβούλευσης και ελπίζουν εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τους στηρίξουμε ιδιαίτερα για να απομακρυνθούν πλήρως τα απόβλητα, να απευθυνθούμε και πάλι στο γαλλικό κράτος, για να τονίσουμε ότι μόνο τα απόβλητα υδραργύρου δεν είναι, να απομακρυνθούν μόνο αυτά δεν είναι συμβατό με την αρχή της πρόληψης και σημαίνει ότι θα υπάρξει κίνδυνος για τον πιο μεγάλο και πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα της Ευρώπης, της κοιλάδας του Ρήνου και γι' αυτό η πλήρης απομάκρυνση θα είναι η μόνη λύση που διατηρεί τον υδροφόρο ορίζοντα. Είναι ακριβή λύση, αλλά πώς θα μας κοστίσει μία ανεπίστρεπτη μόλυνση. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω η Επιτροπή μας πρώτον να επιμείνουμε και πάλι, να επιμείνει και πάλι έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνει ε, πιο προωθημένες έρευνες για τους πραγματικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, που είναι μάλιστα και διαμεθοριακοί, λόγω αυτού του χώρου απόθεση στην Αλσατία. Η Επιτροπή μας λοιπόν, βεβαίως αυτό που προτείνω δεν συμβαίνει συχνά, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό για να είναι σωστή λύση, να απευθυνθούμε απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος και να του ζητήσουμε άλλη μια φορά να εξετάσει το ενδεχόμενο πλήρησης του χώρου στο Καμίν να εξετάσουμε και τη θέση της επιχείρησης ίσως θα είχε έννοια η Επιτροπή μας να τον καλέσει και εκείνον να αναλάβει περισσότερο τις ευθύνες του για το περιβάλλον και να αντιμετωπίσει σοβαρά το ενδεχόμενο της πλήρους απομάκρυνσης αυτού του χώρου απόθεσης. Γιατί υπενθυμίζω ότι αυτό ε, και ιδίως η φύση των αποβλήτων που έχουν αποτεθεί αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, καταλάβατε ότι ήρθα αλλά βλέπω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει να πει τίποτα γι' αυτό. Θέλει κανείς άλλο το λόγο υπ' αυτού. Όχι. Ωραία. Εάν συμφωνείτε θα την κρατήσουμε ανοιχτή με την πρόταση που έκανε η κυρία Μπελιά. Εντάξει, να γραφούν στα πρακτικά αυτά. Η επόμενη είναι θέμα 21. Μέθοδοι εργασίας της Επιτροπής Αναφορών. Επ' αυτού θα δώσω το λόγο απευθείας σε όσους θέλουν να παρέμβουν για το θέμα αυτό και μετά θα κάνουμε συζήτηση. Ποιος θα ήθελε το λόγο για τις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής μας. Η Μάργαρετ η Μάργαρετ ε, πρώτη θα πάρει το λόγο και μετά ο Πίτερ. Θα το κάνω στα αγγλικά, αν και έχω αποφασίσει να μιλήσω περισσότερα δανέζικα. Αλλά σήμερα θα μιλήσω στα αγγλικά. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για, για την ε, προσπάθεια και για τις συστάσεις, για το έργο. Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πολύ περισσότερες αναφορές αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία, αλλά μπορεί και να μας πνίξει κατά κάποιον τρόπο ε, ως Επιτροπή αυτή η επιτυχία μας, διότι δεν έχουμε τα μέσα για να ανταποκρινόμαστε. Και είναι σαφές, το είπε και η Γραμματεία, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους στη γραμματεία ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους και αυτό πρέπει να είναι σαφές δεν μπορείς να λες στους πολίτες στην Ευρώπη ότι ε, είναι καλοδεχούμενοι να υποβάλουν αναφορές και στη συνέχεια εμείς να τις χειριζόμαστε δίκαια αν τελικά περιορίζουμε εμείς τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα και για το νέο Ευρωκοινοβούλιο ε, πρέπει να έχει Επίγνωστο νέο κοινοβούλιο για το γεγονός αυτό και εξ όσων γνωρίζω είμαστε η μόνη επιτροπή που δεν είχε πρόσθετους πόρους σε αντίθεση με όλες τις άλλες επιτροπές. Και εμείς είμαστε οι εγκύτετοι στους πολίτες επιτροπή και ε, δεν είναι ειλικρινές. Ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να κατηγορούμε τους αυτούς μας ή να πρέπει να, να βρούμε έξυπνες μεθόδους για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Η διαχείριση των αναφορών είναι κρίσιμο ζήτημα για τις εργασίες μας. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο μήνυμα που θα αποστείλουμε στη νέα Επιτροπή. Ορισμένες φορές νομίζω ότι ε, ε, αν ανακαλύψουν την επιτροπή αυτή στις βόρειες χώρες, στη Δανία, στη Φιλανδία, πολλές φορές ε, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα. Αλλά φανταστείτε να την ανακαλύψουν και είναι ενεργοί πολίτες οι πολίτες των χωρών αυτών. Και όπως έχουμε πει και πολλές φορές, ότι πολλές αναφορές οι αναφορές ε, καταδεικνύουν το γεγονό ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά μπορεί να καταδεικνύουν και το γεγονό ότι έχουμε ενεργούς πολίτε. Οπότε πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στα καθήκοντα τη Επιτροπή αυτή. Ε, Ο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τα ζητήματα στα οποία συμφωνούμε. Ε, συμφωνούμε ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι εκείνη η Επιτροπή που έχει την καλύτερη, την πιο άμεση σχέση, σύνδεση με τους πολίτες. Από αυτή την άποψη ε, η Επιτροπή Αναφορών είναι και το, το, ε, το εμβληματικότερο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες. Οπότε το πώς χειριζόμαστε τις αναφορές, τους αναφέροντες Αυτά ε, αντικατοπτρίζουν και τον τρόπο εργασίας του Κοινοβουλίου. Πολλές φορές η ιδιότητά μας αυτή δεν είναι γνωστή σε άλλες επιτροπές αν δεν λάβουμε υπόψη μας και τις ηλεκτρονικές αναφορές, ναι, χρειαζόμαστε, περισσότερες, ε, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, αλλά χρειαζόμαστε και οι κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν και για μας. Κάποιες ε, φορές ε, εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε προβλήματα, δεν είναι πρόβλημα της γραμματείας και ε, να επισημάνω και κάτι ακόμη χρειαζόμαστε την, ε, τις, τις αναφορές, ε, που, αυτές που ε, ε εξετάζουμε εδώ στις συνεδριάσεις μας, είναι οι αναφορές για τις οποίες προσκαλούμε και τους αναφέροντες, όπου διοργανώνουμε συζητήσεις που πολλές φορές μένουν και ανοιχτές γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Κάποιες φορές Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι στις εργασίες μας. Είναι και αυτό ένα, ε, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Ε, ότι θα πρέπει δηλαδή να, ε, να υπάρχουν και αναφορές, να, να υπάρχει και δυνατότητα ε, να χειριζόμαστε αναφορές ε, και να, να δίνονται κάποιες ε, επιπλέον πληροφορίες. Ε, το γεγονός δηλαδή ότι, ε, ε, ότι κάποιες αναφορές έμειναν για πάρα πολλά χρόνια χωρίς ε, να εξεταστούν ή έμειναν ανοιχτές. Αυτό πολλές φορές είναι και δικό μας πρόβλημα και γι' αυτό για όλους αυτούς τους λόγους θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για το έγγραφο αυτό και ταυτόχρονα να πω ε, να προτείνω κάποιες ε, προτάσεις για να καταγραφούν και στα πρακτικά που νομίζω ότι δεν είναι και ιδιαίτερα ριζοσπαστικές απλά ε, αποσαφηνίζουν το έγγραφο της γραμματείας. Το μεγαλύτερο μέρος των επιθυμιών και των προτάσεων αφορά εμάς τους ίδιους, δηλαδή τα, τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Κατά την καταχώρηση, για παράδειγμα, Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι πολλές φορές ε, ε, είμαστε και υπεύθυνοι για την διανομή των επισήμενων αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι το τμήμα ε, καταχώρησης πρέπει βέβαια να γνωρίζει πια αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς ποιες αναφορές δεν καταχωρίζονται θέλουμε να υπάρχουν και κάποιες αναφορές οι οποίες δεν καταχωρίζονται αν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος μέχρι, μέσω αυτού του μηχανισμού. Δεν ισχύει αυτό διότι και αυτές οι αναφορές είναι προσβάσιμες σε μας αλλά μιλώ για αναφορές που δεν είναι στην πραγματικότητα. Αναφορές αυτές δεν χρειάζεται να τις τροφοδοτούμε ε, και να τις διανέμουμε και να ε, σπαταλούμε δηλαδή ώρες εργασίας. Το δεύτερο, όσον αφορά το παραδεκτό, ε, έχω την άποψη ότι τα μέλη εντός δύο μηνών μετά την καταχώρηση θα πρέπει να συντάσσουν έναν να, να λαμβάνουν ένα κατάλογο των αναφορών που θα δείχνει την ημερομηνία καταχώρησης των αναφορών και ε, επίσης, το δικό μας δημοκρατικό δικαίωμα, στη συνέχεια οι συντονιστές θα μπορούν να ε, αποφασίζουν για το παραδεκτό στη βάση, να, ψηφίζουν για το παραδεκτό στη βάση γραπτής ε, διαδικασίας ψηφοφορίας. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό η Γραμματεία μας κάνει μια σύσταση και μετά θα πρέπει ε, εμείς να αποφασίσουμε αν συμφωνούμε με αυτή τη σύσταση, αλλά θα ήταν και καλό επίσης, ενθαρρύνουμε δηλαδή την, τη Γραμματεία, ότι ε, δεν, δεν, δεν, έχει, δεν είναι παραδεκτή ε, μια αναφορά. Αυτό πρέπει να, να μπορούμε να το συζητάμε συναδελφικά αλλά όπως είπα όταν ε, χειριζόμαστε τόσες πολλές αναφορές μέσω του μηχανισμού τότε σπαταλούμε και εμείς πάρα πολλούς, πολλές δυνάμεις και με αποτέλεσμα να περιμένουν για πάρα πολύ καιρό οι αναφέροντες. Δέβη θα στα δώσω όλα αυτά για να τα γράψω, για να τα καταθέσει και στα πρακτικά. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Μία φορά το χρόνο τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να ε, συζητούν με την Κομισιόν τις απόψεις ε, τους ε, όσον αφορά τις παραβιάσεις του άρθρου 258 και 260 του κανονισμού. Καλώς κάνουμε και ε, παραπονούμαστε Ίσως μάλιστα η Κομισιόν ελπίζει κιόλας να ξεχάσουμε κάποιες αναφορές. Εμείς σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε και αυτό είναι και μια κλασική περίπτωση κατά την οποία μπορούμε να ε, αποφασίσουμε να συντάξουμε και μια έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, έχει συμβεί αυτό στο παρελθόν. Τώρα όσον αφορά την κατανομή των εκθέσεων. Λοιπόν τώρα οι αναφορές για τις οποίες έχουμε ζητήσει η γνώμη της Κομισιόν θα πρέπει μέσα σε δύο μήνες να έχουμε αυτή την απάντηση. Στόχος μας πρέπει να είναι αυτός. Όταν έχουμε μία αναφορά και ζητάμε να μας δώσει γνώμη η Κομισιόν και μας το κάνει. Τότε, μέσα σε δύο μήνες, εφόσον έχουμε την απάντηση της Κομισιόν, μπορούμε μετά από ζήτηση στην Επιτροπή μπορούμε είτε να κλείσουμε την αναφορά ή να την αφήσουμε ανοιχτή και να γίνουν οι μεταφράσεις και επίσης να προσθέσω, αν αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, τότε εντός τριών μηνών πρέπει να μπει στην μέση διάταξη. Βεβαίως και εδώ είναι δική μας υποχρέωση αυτή. Εφόσον έχουμε πάρει μια απόφαση, τότε τα μέλη της Επιτροπής μας θα πρέπει να θυμούνται τις αποφάσεις μας. Αφήσαμε ανοιχτή μια αναφορά και καμιά φορά μετά έχω την εντύπωση ότι αρκεί αυτό στα μέλη της Επιτροπής μας και ξεχνάνε την αναφορά. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι σωστή αντιμετώπιση. Κατόπιν ε, σημαντικές οι προθεσμίες. Είχαμε μια θρελική συνεδρία στο Στρασβούργο όπου είχαμε πολύ έντονη ανταλλαγή απόψεων για το τι θα κάνουμε για αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι πρέπει να θέτουμε εμείς τις προθεσμίες μας. Γιατί ισχύουν κυρίως και για μας γιατί ξέρετε και εμείς εμείς θέτουμε τις προθεσμίες και πρέπει να ισχύουν και για μας και όταν ε, συντάσσουμε την ημερήσια διάταξη ως συντονιστές θα πρέπει έξι εβδομάδες πριν να έχουν όλη την πληροφόρηση οι συντονιστές και ο πρόεδρος ξέρω κι εγώ Επίσης ε, πάντα προσκαλούνται οι αναφέροντες με πρόταση των συντονιστών. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την ημερήσια διάταξη και να αποστέλλεται με την συμφωνία του Προέδρου πέντε μέρες πριν τη συνεδρίαση, γιατί και τα μέλη πρέπει να ξέρουν τι θα συζητηθεί στην Επιτροπή. Και επίσης το σχέδιο πρακτικών πρέπει να στέλνεται με τη συμφωνία του Προέδρου τρεις μέρες μετά τη συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεών μας. Επίσης, αν περάσει από β σε α σημείο μία αναφορά, συνήθις διαδικασία, Κάποιος μπορεί να το προτείνει στη γραμματεία. Η γραμματεία κάνει μια πρώτη έκθεση όπου λέει ποιες αναφορές πρέπει να κλείσουν όσοι μια β. Αυτός ο κατάλογος αποστέλλεται στα μέλη και τα μέλη το αργότερο μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση μπορεί να τροποποιηθεί προτάσεις των μελών. Εάν ωστόσο μέλη από δύο πολιτικές ομάδες έχουν αντίρρηση, τότε μπορεί να περάσει σε σημείο α μία αναφορά. Εάν ε, ο αναφέρον ή τα μέλη δεν έχουν πληροφορίες για δύο, για μήνες, τότε κλείνει αναφορά και αυτό δεν είναι παράλογο. Το προτείναμε και την τελευταία φορά στο Στρασβούργο. Το θεωρώ αυτονόητο. Αν υπάρχει θέμα συζήτησης. Ε, Βεβαίω δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αν κάποιο προτείνει να περάσει από Β σε Α, πρέπει να αναφέρει και του λόγου. Γιατί ξέρετε ότι αν όλες γίνονται α, αυτό ε, μπλοκάρει την εξαγωγή των εργασιών μας. Τώρα, κανόνες για τη διαδικασία επίγοντος θα πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Η διαδικασία κατεπήγοντος να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Όπως λέει και το όνομά της ε, επίγουσα διαδικασία. Γιατί αλλιώ γίνεται η κανονική διαδικασία. Και επειδή έχουμε τόσο πολλές αναφορές πρέπει να είναι εξαίρεση η επίγουσα διαδικασία και τα μέλη δεν πρέπει πάνω από 10 τέτοια θέματα να θέτουν. Τώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται αυτός ο αριθμός, δεν ξέρω τι θα πει η Μάργαρετ, γιατί χρειαζόμαστε νούμερα, αλλά νομίζω πως θα ήταν καλό για την Επιτροπή μας και ηρεμή και τη Γραμματεία, αν ξέρουν και εκείνοι ότι είμαστε συγκρατημένοι για τα θέματα αυτά. Το τελευταίο σημείο προκάλεσε και ευθυμία την τελευταία φορά στο Στρασβούργο είναι το πώς θα κλείνουν ε, αυτές οι, οι ωραίες κοιμόμενες. Είναι αυτές οι αναφορές που τα μέλη της Επιτροπής φαίνεται ότι τις έχουν ξεχάσει από προηγούμενες θητείες όπου δεν ε, διαπίστωσε παραβιάσει η Κομισιόν και για τις οποίες για μήνες δεν έχουμε συζητήσει θα έπρεπε λοιπόν κάθε καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, να κλείνουν ως μία Β. Τι σημαίνει αυτό. Ξέρω ότι ορισμένοι συγχύζονται και θεωρούν ότι θέλουν να επιβάλλουν οι μεγάλες ομάδες, ε, στις μικρές ομάδες ε, την άποψή τους, αλλά λέω πριν από κάθε διακοπή το καλοκαίρι να δούμε ποιες αναφορές δεν μπορέσαμε να κλείσουμε μεν, αλλά να προσέχουμε να μην παραμένουν αυτές οι ωραίες κοιμόμενες. Τώρα, σχέση με άλλους θεσμούς. Καλά πάμε. Βεβαίως υπάρχει αυτή η ακρόαση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Κατά τη γνώμη μου, ένα αισιόδοξο θα μπορούσε να πει ότι επιτύχαμε μερικώς. Ο απεσιόδοξος θα έλεγε ότι δεν επιτύχαμε όσα θα θέλαμε η Επιτροπή Αναφορών συμμετέχει με βάση το άρθρο 50 μαζί με τις αρμόδιες επιτροπές στην οργάνωση επιτυχημένων πρωτοβουλειών των πολιτών. Και ποια είναι η αρμόδια επιτροπή καθορίζει η διάσκεψη των Προέδρων. Συνήθως θα πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ούτω ώστε οι αρμοδιότητες που έχουμε λάβει να συνεχίσουν να υπάρχουν κατά τη διαδικασία Κροάσεων για τις ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες των πολιτών. Μέχρι στιγμής ήμασταν η κύρια δύναμη, αλλά τώρα τελευταία έχει αλλάξει λίγο η κατάσταση για τον διαμεσολαβητή. Η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια για τη σχέση με τον ε, διαμεσολαβητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα είμαστε αρμόδιοι ο οποίος διαμεσολαβητής μάλλον είναι αρμόδιος για τις αναφορές των πολιτών για θέματα κακοδίκησης. Η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη και για την εκλογή του διαμεσολαβητή και έχουμε τακτική επαφή. Συνολικά λοιπόν καλά τα πάμε. Τελευταίο. Τελευταίο. Συμπληρωματικές οδηγίες για τις αποστολές ε, εξακρίβωσης καταστάσεων. Fact finding. Πολλά επιτύχαμε τον τελευταίο καιρό σε πολλές τέτοιες αποστολές. Υπήρξε μια καινοτόμα διαδικασία. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτός που προτείνει μια τέτοια αποστολή είναι βέβαια ο πρώτος που συμμετέχει και θα πρέπει να καθορίζονται κατάλληλα και οι άλλοι συμμετέχοντες. Γίνεται συνήθως. Σημαντικό είναι και πάλι είναι έτοιμα προς τα μέλη της Επιτροπής μας το αργότερο τρεις μήνες μετά την αποστολή να έχουμε ένα έγγραφο εργασίας το οποίο να είναι το πολύ 7 σελίδων. Μπορούμε να συζητήσουμε αλλά νομίζω ότι η ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι αποστολέ είναι να διευκρινιστούν κάποιες καταστάσεις. Αλλά δεν βοηθάει όταν αργούν πολύ οι εκθέσει μετά. Έχουμε κάνει αποστολέ και χρειάστηκε ένας χρόνος μέχρι να υπάρξει έκθεση για την αποστολή. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε σε τρει μήνες αυτή την ε, έκθεση. Δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 7 σελίδε, όπω είπα. Και ε, κάτι που επίσης είχαμε συζητήσει και επιμένω και από πλευρά της ομάδας μου πρέπει να έχει δύο τμήματα αυτό το έγγραφο εργασία, ένα περιγραφικό και ένα με πορίσματα. Ο επικεφαλής αντιπροσωπείας πρέπει να κάνει τις συζητήσεις τις προπαρασκευαστικές ή να τις αναθέσει κάποιον άλλον. Είπα λοιπόν ότι το έγγραφο αυτό θα το, δώσω τα θα το δώσω στον David για τα πρακτικά Ας το δούμε τώρα απ' έξω, ως κάποιος που αναφέρει. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις. Όταν μας γράφει ένας αναφέρον, όταν υποβάλλει μία αναφορά, τότε νομίζω ότι κοινός μας στόχος πρέπει να είναι ο εξή. Αν μας τη στέλνει ηλεκτρονικά, βεβαίως έχει αμέσως την επιβεβαίωση. Όταν μας γράψει, βεβαίως πολύ καλά του στέλνουμε μία απάντηση Αγαπητέ αναφέροντα, λάβαμε την αναφορά σας. Το αργότερο που θεωρώ... Ναι, ναι, λειτουργεί το σύστημα, λειτουργεί. Αλλά νομίζω λοιπόν ότι το αργότερο τρεις μήνες μετά θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μάθει αν έγινε παραδεκτή ή όχι η αναφορά του. Και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Το ξαναείπα, πρέπει να ξέρει ο αναφέρον. Θα συνεχίσει να εξετάζεται η αναφορά μου ή θεωρούν ότι πρέπει να επιλέξω άλλη οδό. Αυτά μπορούν να γίνουν πολύ γρήγορα εάν πραγματικά έχουμε καλύτερο τρόπο εργασίας. Όταν έχουμε μία αναφορά, όταν έχουμε και την συμβολή της ε, Κομισιόν, εάν θεωρήσουμε κατόπιν ότι μπορούμε να την κλείσουμε ως σημείο Β, τότε θα κλείσουμε ένα μεγάλο τμήμα των αναφορών. Και για να σας καθησυχάσω, εάν νομίζετε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι πιο γρήγορα. Ξέρω ότι ορισμένες φορές ο αναφέρον δεν είναι ευχαριστημένος. Μάργαρετ, ε, σε σένα μιλάω. Μάργαρετ. Μάργαρετ. Το έθεσα στην εμείς διάταξη για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Κατά λίγο, κατά λίγο. Μα αφού με διέκοψαν. Αλλιώ θα είχα τελειώσει. Λοιπόν, ό,τι και αν το, αν το ανακοινώσουμε, θα πρέπει να έχει στην επιστολή μας ο αναφέρον το δικαίωμα να αντιδράσει. Οπότε έχουμε ένα διάλογο με τον αναφέροντα. Θα δώσω λοιπόν για τα πρακτικά όλα όσα είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή όλων σας. Λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Θα είμαι σύντομη. Ήθελα να μιλήσω εγώ, αν μου το επιτρέπεις. Μάργαρετ, αν θες να, προ... εσύ, έλα εδώ να προδέψεις. Εντάξει. Μα τι Μάργαρετ, ξέρεις τι θα πω από τώρα. Λοιπόν, πρώτον. Ο καθένας παίρνει το λόγο και μιλάει χωρίς να διακόπτεται. Αυτή είναι η πρώτη αρχή ε, όλων των Επιτροπών Μάργαρετ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Πίτερ Γιάρ και τον κύριο Μποστινάρου που δεν είναι παρόν γιατί έκανε μια προσπάθεια. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, εδώ παρουσιάζουμε, παρουσιάζουμε Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει σεβασμός και χρόνος γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους μας το θέμα αυτό να ξέρουμε τι μεθόδους εργασίας θα έχει η Επιτροπή μας. Μπορείτε να διαφωνείτε. Θα πάρεις το λόγο για να το πεις. Όσο χρόνο θέλεις. Αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς που έκαναν την προσπάθεια, που άλλοι δεν την έκαναν, να κάνουν αυτή την εργασία. Άλλοι θα μπορούσαμε να την έχουμε κάνει και δεν την κάναμε. Ευχαριστώ τον κύριο Πέιτερ Γιάρ και τον κύριο Μποστινάρου επίση. Λοιπόν, αν τώρα Μάργαντε θες το λόγο, πάρ το λόγο. Με μικρόφωνο. Κοιτάξτε, τα έχουμε συζητήσει αυτά ξανά και ξανά. Ε, πρέπει να πάρουν αποφάσεις και κάθε φορά που οι αποφάσεις δεν είναι υπέρ του ΕΛΚ τότε ξαναμπαίνει το θέμα στην ημερησία και ξαναμπαίνει και ξαναμπαίνει και ξαναμπαίνει. Δεύτερον, έχουμε κανόνες και δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουν πρόβλημα οι κανόνες. Ποιος ε, ε, διαγράφει τους κανόνες, ποιος αλλάζει την ημερησία διάταξη σχεδόν μια μέρα πριν, εσείς. Εσείς αλλάζετε ξανά και ξανά την ημερησία διάταξη. Και ποιος ε, ακυρώνει τις διερευνητικές αποστολές, εσείς πάλι. Έχετε την πλειοψηφία και ήταν πολύ ουγγρικής, ε, ουγγρικού τύπου η συνεδρίαση στο Στρασβούργο και ε, όταν είχαμε την ε, αποστολή στη Γαλλικία δεν μπήκαμε στον κόπο να δούμε τους κανόνες της πλειοψηφία και κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Το μεταθέτετε, το μεταθέτετε και ενδεχομένως θα ακυρώνετε αν δεν σας συμφέρει. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά το σεβασμό των κανόνων. Έχουμε πέντε χρόνια εμπειρίας, τα είδαμε πέντε χρόνια και είδαμε ε, πολλές φορές να παραβιάζονται οι κανονισμοί. Λέμε πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ε, μεταξύ μας. Ναι, φυσικά συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε ε, και σε πλήρη σεβασμό με τον αναφέροντα και αυτό και με αυτό συμφωνώ. Όλα αυτά είναι προφανή και εγώ θα ήθελα να γίνονται έτσι τα πράγματα αλλά να υπάρχουν κανόνες και λόγοι βάσει των οποίων ε, γίνεται παραδεκτή ή όχι μία αναφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνονται σεβαστά τα συμφωνηθέντα. Και όχι εγώ αποφασίζω γιατί, διαφορετικά γιατί έχω την πλειοψηφία μαζί μου. Κάποιοι από τους κανόνες σας ε, δεν είναι εντάξει, αλλά Εν πάση περιπτώσει το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να παραμένει ε, όπως το έχουμε κανονίσει, το έχουμε ρυθμίσει και θα πρέπει να έχει και τους απαραίτητους πόρους, τα κονδύλια τα οποία ε, χρειάζονται. Ναι, βεβαίως λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, είναι προφανές. Επίσης θα πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες και όχι μονάχα ε, αυτούς που μας βολεύουν ή που έχουμε κάνει μόνοι μας εμείς, αλλά και όλους τους κανονισμούς του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν και τέτοιοι κανονισμοί. Τώρα έχουμε, ε, ε, το, την ηλεκτρονική πύλη και ελπίζω ότι θα το σεβαστείτε αυτό. Δεν είναι δυνατόν και γι' αυτό να αλλάζετε συνέχεια την απόφαση γιατί από εκεί προκύπτουν τα περισσότερα προβλήματα σε αυτήν την Επιτροπή. Στην επόμενη, στο επόμενο Κοινοβούλιο ελπίζω ότι θα, γίνει σεβασμός, θα γίνουν σεβαστές οι αρχές της δημοκρατίας και θα γίνουν σεβαστές και οι απόψεις της μειοψηφίας, γιατί έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ε, λοιπόν, εδώ δεν έχουμε απόφαση ε, ήταν μία ε, μακρά διάλεξη σχετικά με το ποιου κανόνες ε, συμπεριφορά θα πρέπει να ακολουθείτε εσείς, Πίτερ. Και α, καλά είναι που δεν είναι εδώ ο κύριος Μποστινάρου, είχα περισσότερο άχτια με, το, με αυτόν, γιατί βλέπουμε ξανά και ξανά τα ίδια πράγματα και να σας πω ότι νομίζω ότι εάν πάρουμε κάποια απόφαση, αν, κάνουμε, αν αποφασίσουμε να κάνουμε μία διαρευνητική αποστολή, να την ολοκληρώσουμε γιατί ο επικεφαλής αυτής της αποστολής δεν έχει, ε, τις, ε, δεν έχει πλήρες εξουσίες. Αν βρεθεί σε μειοψηφική θέση πρέπει να το δεχτεί. Και ελπίζω ότι είναι η τελευταία φορά που ακούμε ε, αυτά τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας από το ΕΛΚ για το πώς θα έπρεπε να ε, κανονίζονται τα πράγματα και να ρυθμίζονται. Αργά βλέπεις, κανείς δεν σε διακόπτει και μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις. Μπορείς να μιλήσεις, κανείς δεν σε διακόψε. Αλλά σου λέω ότι και εγώ ως μέλος του ΕΛΚ ότι ε, δεν θα κάνεις μαθήματα σε κανένα. Δεν δικαιούσε να κάνεις μαθήματα. Λοιπόν, στη δημοκρατία ο πρώτος κανόνας είναι ότι υπάρχουν μειοψηφίες και, και πλειοψηφίες. Και κοίτα, αν θέλεις να αλλάξει, να είσαι στην πλειοψηφία, να πας να γραφτείς το λαϊκό κόμμα στη χώρα σου, να εκλεγείς με αυτούς και τότε θα ανοίξει την πλειοψηφία. Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει για το θέμα αυτό. Κανείς άλλος. Α, ο Γιάρ. Ο Πέτερ Γιάρ. Ναι, πολύ σύντομα. Μαργαρέτε. Είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τον τρόπο εργασία στο τέλος της νομοθετικής θητείας. Και ήταν καλό αυτό. Γιατί έτσι είπαμε ότι όλοι θα φύγουμε ευχαριστημένοι προς τις εκλογικές μας περιφέρειες και θα επανέλθουν κάποιοι με νέα δύναμη στην Επιτροπή. Κοίταξε Μάγκαρετ. Η ΕΛΚ δεν έχει υποψηφία στην Επιτροπή μας. Δεν έχει πλειοψηφία. Θα μου άρεσε να την είχαμε, αλλά δεν έχουμε. Δεν είναι σωστό λοιπόν να λες ότι αξιοποίησε την πλειοψηφία του του ΕΛΚ. Δεν έχουμε πλειοψηφία. Και δεύτερον, για να λήξουμε με κάτι θετικό τώρα τέλος της θητείας είναι, στην ουσία συμφωνούμε να υπάρχει μια διπλή απόφαση. Οι κανόνες υπάρχουν για όλους. πρέπει να τους θυμόμαστε. Να παίρνουμε μια, είπαμε ότι θα πάρουμε μια διπλή απόφαση. Θέλουμε καλύτερου κανόνες, κανόνες που μας, να μας δεσμεύουν εμά τους ίδιου και δεύτερον, οπωσδήποτε, χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό. Αυτή τη διπλή απόφαση πρέπει οπωσδήποτε να τη δώσουμε στον πρόεδρο της Επιτροπής μας για να επιτύχουμε κάτι. Ε, χαιρόμαστε που έχουμε πολλές ε, αναφορές θέλουμε να υποβάλουν αναφορές οι πολίτες. Τώρα έχουμε και την ηλεκτρονική αναφορά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια διαδικασία που να μας επιτρέπει ως Επιτροπή και η Γραμματεία μας να είμαστε σε θέση σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ανταποκρινόμαστε στην Επιτροπή. Αυτό είναι το πρόβλημα, το κοινό μας καθήκον και μέχρι στιγμής η Επιτροπή Θα πήγε πολύ καλά. Πολύ λίγες ε, ήταν ε, αποφάσεις που βασίζονταν μόνο σε μία ομάδα. περισσότερες ήταν κοινή αποδοχής. Αν απέτυχε μία διερευνητική αποστολή, δεν είναι θέμα του ΕΛΚ. Είναι θέμα του δεν υπήρχαν άτομα που να θέλουν να συμμετάσχουν. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Ο κύριος Φιλίπ Μπουλάουγκ. Ευχαριστώ, Κάρλος. Ήθελα απλώς να απαντήσω σε αυτό που ακούστηκε. Το ΕΛΚ δεν έχει ε, πλειοψηφία και για να βρει την πλειοψηφία κάνει συμμαχίες με άλλες πολιτικές ομάδες. Αυτό είναι ο κανόνας της δημοκρατίας. Δεύτερον, πιστεύω ότι οι προτάσεις που ε, υπευλήθησαν στο έγγραφο αυτό προκύπτουν από διαπιστώσεις που κάναμε στη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής μας ε, και στην ίδια την Επιτροπή αλλά και στη διάρκεια των διερευνητικών αποστολών ε, τις οποίες οργανώσαμε ε, και στη διάρκεια των οποίων εργασιών και αποστολών διαπιστώσαμε ότι ε, το σύστημα δεν λειτουργούσε τέλεια και ότι υπήρχαν ελλείψεις οι οποίες προέκυπταν από αντίστοιχες ελλείψεις των κανονισμών. Ε, γι' αυτό λοιπόν θεωρήσαμε σκόπιμο ε, στο τέλος της θητείας ε, οι απερχόμενοι βουλευτές να κάνουν μια αποθυσάβριση ας πούμε των ε, μαθημάτων ε, και των διδαγμάτων της θητείας τους έτσι ώστε να τα μεταφέρουν στους νέους βουλευτές ε, για να τους ευαισθητοποιήσουν στα προβλήματα αυτά χωρίς όμως να και ταυτόχρονα να προτείνονται κάποιες λύσεις γιατί οι νέοι βουλευτές δεν θα έχουν την απαραίτητη απόσταση ας πούμε έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Δόθηκαν λοιπόν, έγιναν οι συγκεκριμένες προτάσεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ΕΛΚ προσπαθεί να παίξει ηγεμονικό ρόλο, ειδικά δε σε τούτη την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Φιλίπ. Λοιπόν, εδώ στο Προεδρείο έχω τρία έγγραφα. Ένα έγγραφο του των κυρίων Γιάρ και Μποστινάρου, όπως είπα και προηγουμένως. Άλλο, που το εξεπώνησε η Γραμματεία και ένα πιο σύντομο κάποια ανάλυση της κατάστασης που κάνει η Πρόεδρος, η κυρία Ματσόνη. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω, θέλετε να το ψηφίσουμε. Είμαστε 7 τακτικά μέλη. 6-7. Ο κύριος Γιάρ. Στην τελευταία συνεδρία των συντονιστών είχαμε συμφωνήσει ότι η Γραμματεία θα συντάξει ένα έγγραφο εργασίας ε, οι ευρωβουλευτές να υποβάλουν δικές τους προτάσεις αλλά ομόφωνα αποφασίσαμε ότι δεν θα υπήρχε ψηφοφορία και νομίζω ότι πρέπει να την τηρήσουμε αυτή την απόφαση για να μην ε, ε, αξιοποιήσουμε τυχαίου συσχετισμού δύναμη. Άρα ε, να, το, να γραφτεί και στα πρακτικά δεν θα γίνει ψηφοφορία. No vote, Margaret. Βλέπεις ότι ακόμη και στο τέλος της θητείας ε, εμεί σηκώνουμε και μια λευκή σημαία προς την πλευρά σου. Α, δεν το ήξερα. Δεν ήμουν στου συντονιστέ. Ωραία. Άρα όλοι συμφωνούμε. Έγινε αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Ναι, ναι, ο κύριος Βίλαντ. μια ιδέα για το μέλλον. Ξέρω ότι η Γραμματεία έχει πολύ μεγάλο έργο και ιδιαίτερα όσον αφορά τις, νέες, ε, ε, τις εκλογές. Ε, νομίζω πάντως ότι σε άλλα κοινοβούλια όπου υπάρχουν επιτροπές αναφορέων και ενδεχομένως έχουν και υπάρχουν και θετικές εμπειρίες, ίσως θα μπορούσαμε ε, να ζητήσουμε ποιε είναι οι μέθοδοι εργασίας που χρησιμοποιούν εκείνα τα κοινοβούλια, ώστε ε, να εμπλουτίσουμε και εμείς τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ωραία. Λαμβάνουμε υπόψη και τα σχόλια του κ. Βίλαντ και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της μερικής διάταξης η αναφορά 22 κάρτος 2010 του Ματίας ε, Λαμπλάσκο από την ομάδα για ε, την ιστορική μνήμη για να γίνει η 22 Ιουλίου η μέρα μνήμης για τα θύματα εγκλημάτων μίσους. Η κυρία Αντρές ε, θα μιλήσει για το θέμα αυτό εκ μέρους του αναφέροντος. Ευχαριστώ όπως είπατε. Είναι μια αναφορά του κυρίου Ματίας Αλόνσο Μπλάσκο εκ μέρους της ομάδας για την ανάκτηση της ιστορικής μνήμης που ζητάει να υπάρχει μια μέρα μνήμης για τα θύματα μίσους και να είναι 22 Ιουλίου τότε που έγινε αυτή η μαζική δολοφονία στο Όσλο στο νησί Ουτόγια. Να είναι λοιπόν μια μέρα υπέρ της ε, δημοκρατίας, ε, της πολυμορφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το στείλαμε το θέμα αυτό στο Προεδρείο, αλλά δεν έχει υπάρξει απάντηση. Είναι πολύ απλή πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Ανδρέας Μπαρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, δεν είναι κανείς. Α, είναι ένα θέμα πολιτικό. Ωραία. Έχετε δίκιο κυρία Ανδρές Μαρία. Υποθέτω ότι έχετε και την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος Μάρτιν Σούλτς απαντώντας την ερώτηση που του, στην επιστολή που του έστειλε η κυρία Ματσόνη ο πρόεδρος όπως μας είπε ότι απέστειλε το θέμα αυτό στη διάσκεψη των προέδρων αλλά το ότι δεν υπήρξε καμία απάντηση από τους ε, προέδρους των πολιτικών ομάδων. Άρα νομίζω ότι θα έπρεπε να απευθυνθούμε και πάλι στον κύριο Σούλτς και τη διάσκεψη των προέδρων, εφόσον είναι αρμόδιοι γι' αυτό, να μας πούν ποια είναι η άποψή τους. Εντάξει. Ναι, ναι, πολύ σωστό. Και καλό θα ήταν η Επιτροπή Αναφορών να καθορίσει επίσης τη θέση της για αυτήν την θέση του αναφέροντος, την πρόταση του αναφέροντος. Δηλαδή να στηρίξουμε αυτή την ιδέα έναντι της Επιτροπής των Προέδρων, της Διάσκεψης των Προέδρων. Εντάξει, πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Έτσι θα το κάνουμε. Το επόμενο θέμα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Φτάσαμε σε συμφωνία σήμερα το πρωί να βάλουμε κάτι για το Ίδρυμα Νεότητας, Jugendamt. Έχω ένα κατάλογο αναφερόντων, έξι είναι, τους οποίους καλωσορίζω στην Επιτροπή Αναφορών. Το μόνο που θα σας παρακαλούσα είναι υποθέτω ότι θέλουν να μιλήσουν και οι έξι. Παρακαλώ, έχουμε περιορισμένο χρόνο. Θα δώσουμε τρία λεπτά στον καθένα. Δεν θα έχετε 18 λεπτά συνολικά. Συνήθως μία αναφορά μας απασχολεί 5-6 λεπτά. Όχι, λέει μια κυρία, δεν συμφωνεί. δεν είναι δυνατόν μετά από τέσσερα χρόνια που περιμένουμε να συζητηθούν οι αναφορές μας αφού έχουν μπει πλέον στη μερίσια διάταξη ε, να ε, έχουν διαγραφεί ε, έτσι ώστε να μην μπορούν να έρθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και μετά από τόσο καιρό να ξαναμπαίνει ξαφνικά στη μερίσια διάταξη και να έχουμε τρία λεπτά ο καθένας. Καταλαβαίνω το σχόλιο σας, αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε στις 6.30, στις 18 και 30. Παρακαλώ, σας άκουσα, παρακαλώ, βάλτε τα ακουστικά σας. Στις 6.30 οι συνεδρίες πρέπει να τελειώσει, γιατί αυτές οι κυρίες και οι κύριοι πρέπει να φύγουν. Τελειώνει το ωράριο εργασία τους. Θέλετε να ξεκινήσει μια συζήτηση. Βεβαίως, πρέπει να μιλήσετε εσείς, η πολιτική, η κομισιόν κτλ. Μια συζήτηση δεν είναι μόνο να μιλήσετε εσείς. Υποθέτω ότι θέλετε να κάνετε ανταλλαγή απόψεων μαζί μας. Οπότε, εάν όλοι θέλετε να μπορέσουν να, μπορέσουν να πάρουν όλοι τον λόγο και λογικό μετά από τέσσερα χρόνια όπως είδατε και άλλες ε, αναφορές καθυστέρησαν και τους δόθηκε πολύ λιγότερος χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν θα περιορίσω τις παρεμβάσεις και των 6 3 λεπτά. Θα μπορώ να σας δώσω 4 στον καθένα. Αυτό θα έκανε 24-25 λεπτά που θα παρέμβετε εσείς. Σας διαβεβαιώ ότι κανένας δεν λαμβάνει για να παρουσιάσει θέμα 25 λεπτά. Οπότε θα σας παρακαλούσα να είστε συγκεκριμένοι, 4 λεπτά ο καθένας και μετά να έχουμε τη συζήτηση μεταξύ όλων μας. Γιατί νομίζω ότι θέλετε να ε, γίνει συζήτηση. Ναι, αν μπορέσουμε να απαντήσουμε, βεβαίως. βεβαίως. Λοιπόν, θα πάρετε πρώτο λόγο. Μετά θα παρεύει κάποιο από την Επιτροπή. Δεν έκανε την Επιτροπή. Α, ωραία. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στα αιτήματά σα. Κυρίως είδαμε ότι και ότι μόλις έφυγε και ο Ευρωβουλευτής, Γερμανός Ευρωβουλευτής, ο οποίος ε, ζήτησε να μην εγγραφεί το θέμα στη Μέση Διάταξη. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, ο κανόνας είναι. Εισάγουν το θέμα οι αναφέροντες, ε, απαντάει η Κομισιόν και μετά γίνεται μια ζήτηση μεταξύ των βουλευτών ε, και μπορείτε και εσείς να παρέμβετε. Σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχει κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είναι θέμα δική μα ευθύνη η γραμματεία, διότι αυτό που μου υπόθηκε είναι ότι αποφασίστηκε σήμερα το πρωί να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Εντάξει, με βάση αυτέ τι συνθήκε θέλετε να παρουσιάσετε το θέμα. Τι σημαίνει εάν, εάν συζητήσουμε τώρα δεν θα απαντηθεί το θέμα μας όχι γιατί δεν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε τι θα συζητήσουμε. Δηλαδή ποια μπορεί να είναι η λύση ας πούμε, ποια μπορεί να είναι η συνέχεια της καταστάσεως. Εμείς μπορούμε να, ε, θέλουμε να καταλάβουμε τι γίνεται, εμείς να σας εξηγήσουμε πώς έχουν τα πράγματα, αλλά δεν θα πάρουμε καμία απάντηση, αυτό θέλετε να μου πείτε. Κοιτάξτε λυπάμαι ιδιαίτερα, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, το παραδέχομαι. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση και αυτή την απάντηση να γίνει συζήτηση μεταξύ ε, ημών και των βουλευτών. Αλλά ο κύριος Μπουρλάν θέλει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Νομίζω ότι λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση η οποία είναι ιδιάζουσα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είναι εδώ, θα έπρεπε η Επιτροπή να περιμένει την απόφαση ε, που θα έπαιρνε σήμερα το πρωί η Επιτροπή μα ε, για να αποφασίσει αν θα στείλει κάποιον. Επομένω, ένα δίκο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Έγινε μια προσπάθεια να ε, βγει το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεγονό ότι τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ελαμβάνεται 9 η ώρα το πρωί κατά τη συζήτηση ε, του περιεχομένου της ημερησίας διατάξεως. Ευρωμένως η Κομισιόν έπρεπε να περιμένει ποια θα ήταν η απόφασή μας 9 η ώρα το πρωί για να ε, στείλει τον ε, εκπρόσωπό της. Επομένως δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, είναι εκείνη ένα δίκο. Δεν είναι πρόβλημα των αναφερόντων. Οι αναφέροντες είναι εδώ, επομένως πρέπει να πάρουν το λόγο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας στείλει απαντήσεις γραπτά. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι, βεβαίως και για σεβασμό από τους, ε, για τους αναφέροντες που έρχονται από τόσο μακρά, μακριά θα ανοίξω τη συζήτηση, αλλά δεν μπορεί να γίνεται έτσι μια συζήτηση. Μια συζήτηση χωρίς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες μας. Αλλά εάν δεν έχετε πρόβλημα, σας θέτω το ερώτημα, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους αναφερόμενους. Μπουρλάκη Θεραβέτια. Αλλά θα πρέπει να ακούσουμε τους αναφέροντες. Να σας πω την αλήθεια, θα έπρεπε ε, να μην πούμε, να μην ειδοποιήσουμε τους, ε, αναφέρον, αναφέροντες ε, για την διαγραφή μέχρι σήμερα το πρωί που θα ελαμβάνω το η τελική απόφαση. il la réponse.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 Uh, Ζητώ συγγνώμη γιατί η γραμματεία ε, ε, μπαίνει στην συζήτηση αυτή. Ε, είχε ληφθεί απόφαση να μην μπει το θέμα αυτό στη μέση διάταξη. Οι συντονιστές όμως, οι συντονιστές λοιπόν ενέκριναν τη μέση διάταξη χωρίς το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ έγιναν κάποιες συζητήσεις σήμερα το πρωί σχετικά με τα θέματα τα οποία θα μπαίνουν στη μέση διάταξη. Κύριε Μπουρλάντ, κάνατε σήμερα το πρωί μια πρόταση έτσι ώστε να μπει το θέμα στη μέση διάταξη και είχατε και τη στήριξη της πλειοψηφίας της Επιτροπής. Γι' αυτό ακριβώς συμπεριλαμβάνεται το θέμα αυτό τελικά στη μέση διάταξη. Αλλά επειδή ήταν τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση αυτή, δεν υπήρχε η δυνατότητα να ληφθούν οι περαιτέρω, ε, ε, ε τα περαιτέρω μέτρα. Ε, θα έχουν τη δυνατότητα λόγω τη της δικής σας παρέμβασης να μιλήσουν οι, αναφέροντε αναφέροντες ε, και να εκφράσουν την άποψή τους χωρίς να είναι εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόεδρος. Λοιπόν, παρά τις εξηγήσεις η κατάσταση δεν είναι ομαλή. Αλλά εφόσον έχουμε περισσότερο χρόνο, πέντε λεπτά ο καθένας, οπότε μισή ώρα όλοι σας. Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Ποιος θα μιλήσει πρώτος? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ έχω ένα κατάλογο ομιλητών. Πρώτο είναι ο Λαϊπέρνη Πορών Χριστίδη Κολόμπο Ιτζόλη. Ποιο θα είναι ο πρώτο. Ποιο θα πάρει πρώτο το λόγο. Οκ, okay, Κολόμπο θα μιλήσει πρώτη. Παρακαλώ, κύριε Κολόμπο λοιπόν. Eh, Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι το πρόβλημα δεν είναι το Jugendamt της Γερμανίας, αλλά η στάση της Γερμανίας. Ε, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, με αυτές τις αναφορές, με τις επιτροπές που δεν έρχονται, με τον Ευρωβουλευτή που, όταν, ε, που, που δεν ήμουν, όταν δεν ήμουν εδώ, ε, με χαρακτήρισε εγκληματία και τελικά τώρα που είμαι εδώ μπροστά μου δεν λέει τίποτα και έφυγε. Όσον αφορά τώρα τις ε, αναφορές ε, κατά ε, των υπηρεσιών της κοινωνικών υπηρεσιών της Αγγλίας και της Δανίας είχαμε ένα ολόκληρο σοου από πλευρά των Γερμανών και Αυστριακών Ευρωβουλευτών γιατί εδώ αφορούσε το θέμα εσωτερικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο κτλ. Βροντοφώναξαν ότι πρόκειται για οικογενειακά δικαιώματα ε, γιατί ε, σε εκείνη την περίπτωση ήταν δύο ε, παιδιά αυστριακής υπηκότητας τα οποία βρίσκονταν στην Δανία. Αλλά οτιδήποτε ξεπερνάει τα σύνορα της Γερμανίας και της Αυστρίας δεν μπορεί να συζητηθεί. Αυτό ήταν και η μοίρα των δικών μας αναφορών. Εμφανίζονται στην ημερησιαδέτηξη, εξαφανίζονται, συζητιούνται, δεν συζητιούνται κτλ. Ξεκινήσαμε ήδη από το 2009. Το 2010 συζητήθηκε για πρώτη φορά ε, και εκεί διαπιστώθηκε σημαντική παραβίαση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά σιωπή. Εν συνόψη να σας πω ότι έχουμε γερμανό γονέα που δεν ε, μπορεί να ζητήσει τον επαναπατρισμό των παιδιών αλλά όπως πάντα οι γερμανικές αρχές του δίνουν ε, τα έγγραφα τα απαραίτητα. Στη δική μου περίπτωση υπάρχει πλαστογραφημένη μετάφραση ε, και αυτό το έχει πιστοποιήσει η αρμόδια αρχή της Ιταλικής Δημοκρατίας. Και ξέρετε ότι ο άπαξ και κάποιος περάσει τα σύνορα της Γερμανίας δεν ξαναφεύγει ποτέ. αρνήθηκαν στην προκείμενη περίπτωση το δικαίωμα που έχουν οι δύο γονείς με δύο διαφορετικές γλώσσες. Και πρέπει να σας πω ότι ε, σύμφωνα με την επιστολή που πήραμε ε, το, ε, μας αναφέρεται το άρθρο 24 του χάρτη θερμιολόδων δικαιωμάτων δεν εφαρμόζεται πάντα και ότι αν δεν εφαρμόσει τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 24 η Γερμανία δεν παραβιάζει νοσιακό δίκαιο. τελευταία συζήτηση λοιπόν της αναφοράς μου ήταν το 2010. Από τότε δεν ξαναείδα τα παιδιά μου. Με χαρακτήρισαν τρελή, εγκληματία και εδώ βεβαίως, ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με χαρακτήρισαν έτσι οι Γερμανοί ε, βουλευτές, τη απουσία μου φυσικά. Ε, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, έγραψα ένα πρώτο βιβλίο, τώρα ετοιμάζομαι να γράψω ένα δεύτερο παιδί, ε, συγγνώμη ένα δεύτερο βιβλίο, αλλά τα παιδιά μου δεν τα έχω ξαναδεί. έχω είμαι μια γυναίκα λοιπόν ένας γονιός ο οποίος ε, έχει τα μυαλά του για να κάνει ένα σωρό πράγματα αλλά όχι για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. η κατάστασή μου δεν ενδιαφέρει απολύτως κανέναν. οι γερμανικές αρχές ακολουθούν τις δικές τους ε, αποφάσεις. Ε, μου έχουν απαντήσει οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ότι είναι δικιά τους υποχρέωση να κρατήσουν τα παιδιά στην γερμανία και πρέπει να να πω ότι πίσω από αυτή τη στάση υπάρχουν, ε, υπάρχει ένας χορός εκατομμυρίων. Ε, ε, να σας πω επίσης ότι εγώ χάνω το σπίτι το οποίο αγόρασα 12 χρόνια πριν το γάμο μου, χάνω επίσης τις καταθέσεις μου. τώρα τι να σας πω, αν αυτό δεν είναι χορός εκατομμυρίων και μια φάμπρικα που βγάζει χρήματα, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε φορά οι αναφορές οι οποίε είναι πολύ περισσότερε από τι 6 ή 24 ε, οι οποίε είχαν προβλεφθεί αρχικά. Κάθε φορά λοιπόν οι αναφορές κατά της Γερμανίας τελικά δεν γίνονται ποτέ παραδεκτές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι και πρέπει να σας πω ότι τώρα και εν ώψη ευρωπαϊκών εκλογών τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ε, ε, πίσω από κάθε άνθρωπο ε, και κάθε αναφέροντα υπάρχουν φίλοι, οικογένειες, πολλοί κόσμος και αυτοί οι άνθρωποι έχουν πια μπουχτίσει από αυτή την κατάσταση και από τα αντιγερμανικά αισθήματα τα οποία καλλιεργούν οι ίδιοι οι Γερμανοί. Τα παιδιά μας, τα παιδιά μας όταν είτε δεν έχουν γερμανική γερμανική υπηκότητα ή ακόμα χειρότερα μόνο από τον ένα γονιό έχουν γερμανική ή αυστριακή υπηκότητα ε, ξέρουμε ότι ε, δεν έχουν πλέον καμία επαφή με τον άλλο γονιό που δεν είναι Γερμανός ή Αυστριακός και δεν λαμβάνονται υπόψη ε, τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεύτερος ποιος είναι. Να ακολουθήσω τον κατάλογο. Ο κύριος Ζιλμπέρτη. Κύριο Ζιλμπέρτη. Πέντε λεπτά κι εσείς κύριε Ζιλμπέρτη. Με μικρόφωνο. Έβαλα μία αναφορά για την καταχρηστική χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης στα πλαίσια του οικογενειακού δικαίου. Φυλακίστηκα τον Οκτώβριο του 2012 με γερμανικό ένταλμα σύλληψης που συντάχθηκε από το δικαστήριο του Λάνσχουτ που με κατηγορούσε ότι δεν πλήρωνα τη διατροφή μου. Το οποίο ισχύει. Αρνούμε να πληρώσω διατροφή γιατί στην ουσία πρόκειται για λίτρα για τα παιδιά μου διότι το δικαστήριο του Λάνσχουτ και η κοινωνική λειτουργή του Ιδρύματος για την Νεότητα του Λάνσχουτ και η αστυνομία του Λάνσχουτ με αντιμετώπισαν ε, με διακρίσεις, με εξευτέλισαν, με απαγορεύουν να βλέπω τα παιδιά μου, απαγορεύω στα παιδιά μου να έρθουν στη Γαλλία να δουν τη γαλλική τους οικογένεια. Οπότε στις 8 Οκτωβρίου του 2010 έκανα μία απεργία ε, πείνας και δίψας 10 μέρες. Ε, για ένα χρόνο ήμουν από αυστηρό γαλλικό δικαστικό έλεγχο και εκδόθηκα τον Οκτώβριο του 2013 ενώ το δικαστήριο του Λάνσχουτ ήξερε ότι ήταν απαράδεκτο το ένταλμα σύλληψης διότι περιείχε ένα τυπικό σφάλμα ήταν γιατί δεν είχα παραστεί σε ένα δικαστήριο ενώ ε, το κλήτευμα, η κλήτευση είχε σταλεί σε λάθος διεύθυνση. Έδωσα δημοσιότητα στην περίπτωσή μου γιατί νομίζω ότι είναι σκανδαλώδης. Πέρα από τις απειλές ε, που, των οποίων ήμουν θύμα από τη γερμανική αστυνομία πέρα από την παρακολούθηση των ε, τηλεφωνημάτων μου που έγιναν από εισαγγελέα του μονάχου και που αφορούσαν ε, επικοινωνίες με άλλες χώρες, την Ιταλία, την ε, Ελλάδα. Εστάλιν στη Γερμανία, έκανα τουρισμό φυλακών, πήγα σε έξι φυλακές σε δέκα μέρες, βγήκα από τη φυλακή και τώρα θα χάσω τη δουλειά μου. Η απόφαση για την πληρωμή διατροφής δεν έχει καμία νομική ισχύ, δεν είχα υπόψη αυτή την απόφαση, πλήρωνα υπερβολικά διατροφή σε σχέση με την απόφαση της δικαιοσύνης, πλήρωνα 500 με 600 ευρώ το μήνα, ενώ το δικαστήριο ε, είχε επιδικάσει 326 ευρώ διατροφή και όταν διαπίστωσε ότι η πρώην γυναίκα μου ήταν φίλη του δικαστή του Λάνσκουτ και ήξερε όλη τη συμμορία. Και ότι επίσης ε, υπήρχαν σχέσεις με την οργάνωση βοήθεια στην νεότητα που ασχολείται με περιφερειακή βοήθεια προς την νεότητα. Όταν διαπίστωσα ότι ο δικηγόρος ε, της πρώην γυναίκας μου είναι χορηγός αυτής της οργάνωσης όταν διαπίστωσα ότι αντιμετώπιζα μια ολόκληρη ομάδα φίλων που ασχολούνται με την νεότητα αποφάσισα να σταματήσω να πληρώνω διατροφή και είπα στους υπευθύνου ότι επειδή δεν ξέρω πού μένουν τα παιδιά μου δεν ξέρω καν είναι ζωντανά θα σταματήσω να πληρώνω διατροφή. Και η απάντηση των κοινωνικών λειτουργών του Ιδρύματος για την Νεότητα ήταν ότι εφόσον δεν έχω λάβει ληξιαρχική πράξη θανάτου των παιδιών μου πρέπει να πληρώνω. Εντάξει, πολλά μπορούμε να πούμε για το πόσο φροντίζει τα παιδιά η Γερμανία, αλλά αντιμετωπίστηκα με λάθος τρόπο, εξευτελίστηκα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε με την αναφορά μου, γιατί λείπουν διάφοροι, αλλά είναι γεγονός ότι έχω τώρα γαλλική οικογένεια που είναι, αρχι... που είναι... έχω ε, συγγενείς στη Βελγία, στην... Ε, στο Βέλγιο, στην Ιταλία. Δεν είμαι πολύ της δεύτερης κατηγορίας, όπως θεωρούν ορισμένοι κοινωνικοί λειτουργοί στην ε, Γερμανία. Και είναι σαφές ότι θα ξαναμπώ φυλακή για το δεύτερο ένταλμα σύλληψης, το ευρωπαϊκό, γιατί τώρα ο δικαστής Ζούτνερ είπε ότι δεν θα κάνει λάθος, με απειλή ένας δικαστής και όσο δεν θα μπορούν να έρθουν τα παιδιά μου για διακοπές, για να έχω το δικαίωμα επίσκεψη, που είναι απόλυτα σύνηθε στην Ευρώπη, δεν θα πληρώσω διατροφή. Θα είμαι εγκληματίας, όπως λένε διάφοροι πρωταγωνιστές αυτού του έργου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε. Ο επόμενος, Σεντρίκ Λογό. Θα πάρω το λόγο εξ ονόματος ε, του Σεντρίκ Λοχόν, γιατί πρόκειται για την αναφορά Weissenstadt. Ε, ε, και, και στη δική του περίπτωση έχει πρόβλημα σχετικά με αυτό το αίτημα αρρωγής ε, και όπως είναι άλλωστε και η περίπτωση ε, όλων των παρισταμένων ε, γιατί οι Γερμανοί προσπαθούν να περάσουν αυτό το εναλλακτικό μέτρο σαν μέτρο με νομική ισχύ. Θα σας εξηγήσω λοιπόν την κατάσταση του κυρίου Λοραό για τον οποίο υπάρχει μια γαλλική απόφαση της γαλλικής νομοθεσίας βάσει του κανονισμού 39 Βρυξέλλες 2α μόλις ανακάλυψε ότι χρωστάει 6.000 ευρώ ε, ε, στη, στο γερμανικό κράτος γιατί η, η, του σε συνεργασία με την γαλλική ε, σε, συνεργασία με, την γερμανική, με τις γερμανικές αρχές παίρνει αυτό το επίδομα τα τελευταία χρόνια. Βεβαίω εδώ έχουμε μια καταχρηστική κατάσταση, έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν συνάδει δηλαδή με την ελεύθερη και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Θα μπορούσα να σας διαβάσω όλα τα νομικά ε, κείμενα, τα συναφή κείμενα, αλλά νομίζω ότι έχετε ε, την αναφορά ε, μπροστά σας. Ναι, μπορείτε να μας δώσετε, λέει ο Πρόεδρος, αυτήν την αναφορά. Ε, ναι, είναι αναφορά που την έχετε ήδη στα χέρια σας. Ναι, αλλά θα τη βάλουμε να μας τη δώσετε έτσι ώστε να τη βάλουμε στα πρακτικά. Ε, της ε, επιτροπή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο Μιλτή, να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα νομικής προσφυγής γιατί πρόκειται για ένα διοικητικό μέτρο ε, που όμως βάσει του κανονισμού Βρυξέλλες 2α οι γερμανικές αρχές το επιβάλλουν σε ολόκληρη την ενωσιακή επικράτεια. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν την κατάσταση του κυρίου Λωράου ο οποίος μετά από ε, πριν από δύο εβδομάδες κατάλαβε ότι έχει 6.000 ε, ευρώ καθυστερούμενα. εγώ ποιος ξέρει πόσα χρωστάω δηλαδή με αυτόν τον υπολογισμό, ενώ έχω χάσει τα πάντα, τη δουλειά μου, την ιδιοκτησία μου. Στη Γερμανία μου τα έκλεψαν όλα, μου τα πήραν όλα καταχρηστικά. Ξέρετε, στη Γερμανία όταν κανείς δεν μιλάει τη γλώσσα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. παίρνει έναν Γερμανό ε, ε, δικηγόρο ε, στον οποίο δεν μπορεί να έχει καν εμπιστοσύνη γιατί αυτός ο δικηγόρος οπωσδήποτε θα προσπαθήσει να καλύψει την πλευρά των γερμανικών αρχών προς ζημία του πελάτου του. Αλλά είμαστε στην Ευρώπη κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω πολύ σοβαρά προβλήματα με τη Γερμανία, αλλά δεν τα δημιούργησα εγώ ε, το προβλήματα. Κύριε Βίλαντ, οι δικές σας αρχές ε, δημιούργησαν ε, τα προβλήματα αυτά. Τι να σας πω, θα με ρωτήσετε, είμαι γερμανόφοβος, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα έχω μεγάλο πρόβλημα με τη Γερμανία. Έμαθα τη γλώσσα, έμαθα τον πολιτισμό, την κουλτούρα αυτή τη χώρα. Προσπάθησα να αντιμετωπίσω αυτήν τη διγλωσία που έχετε σε νομικό επίπεδο. Έκανα τα πάντα αλλά τελικά μου φερθήκατε σαν να είμαι πολίτης δεύτερης ε, κατηγορίας. Θεωρείτε ότι είμαι εγκληματίας, αλλά εγώ είμαι περήφανος που είμαι τέτοιος ε, εγκληματίας, ε, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένα παιδί πρέπει να έχει τους δύο του γονείς, είτε είναι Γάλλοι, είτε είναι Ισπανοί, είτε είναι οποιασδήποτε ηθαγένειας. Εμείς είμαστε εδώ για να φτιάξουμε την Ευρώπη των λαών και όχι την Ευρώπη της Γερμανίας. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Τόμας Μπρόνκα. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Με μικρόφωνο. Ο κύριος Πουτίν, ο οποίος είναι εδώ και ο οποίος είχε μία σχετική ε, αναφορά, δεν έχει ε, εγγραφεί στον κατάλογό σας. Έχει όμως και αυτός αναφορά σχετικά με αυτό το επίδομα. Στη δικιά του, ε, απλώς ήθελα για να κλείσουμε το θέμα Bisonshaft για να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τον Bison και να μην το ξανασυζητήσουμε. Έλειπε αυτό το, αυτή η ψηφίδα. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Έχω ένα κατάλογο όμως. Ναι, απλώς έλεγα ότι μια και είχαμε τα πέντε λεπτά και είχε προβληθεί το θέμα, είχαν προβληθεί πέντε λεπτά. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά και εγώ είμαι Ευρωπαίος πολίτης, ε. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, λέει ο Πρόεδρος, ε, αλλά υπάρχουν και άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες ε, οι οποίοι είχαν εγγραφεί για να μιλήσουν πριν από εσά. Ο κύριος Τόμας Μπρόγκα δεν είναι εδώ. Α, είστε εδώ. Ωραία, ωραία. Κύριε Μπρόγκ, παρακαλώ. Κύριε και κύριοι, θα σας μιλήσω στα γαλλικά γιατί είναι η γλώσσα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και σας μιλάω για ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2007 με πικρία διαπιστώνω ότι οι γερμανικές αρχές δίνουν ε, ατελείς ακόμα και ψευδείς απαντήσεις όπως έχουν δώσει και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών άλλωστε. Έχω εδώ στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την καθημερινότητα ε, των ε, θυμάτων της γερμανικής δικαιοσύνης. Ε, σας λένε ότι το Ίδρυμα Νεότητας ε, είναι σύνομο, αλλά σύμφωνα με ποιο νόμο. Ε, στην ουσία ψεύδονται όσοι εμφανίζονται ενώπιον των δικαστηρίων. Επίσης δεν υπάρχει καμία διαδικαστική επαλήθευση. Το Ίδρυμα Νεότητας ακυρώνει πραγματογνωμοσύνες ψυχιάτρων, γιατρών που δείχνουν οποιοδήποτε κίνδυνο για τα παιδιά. Δεν εμφανίζονται και δεν γίνονται αποδεκτά τα στοιχεία αυτά από το δικαστήριο τελεία και παύλα. Επίσης ε, ε, σας λένε ότι μπορείτε να επαληθεύσετε ε, τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Νεότητας με προσφυγή στην δικαιοσύνη. Αυτό είναι ψέμα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προσφυγής και δεν αναφέρομαι σε μία μεμονωμένη περίπτωση. Ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Δεν μπορείτε να κάνετε μήνυση ενώπιον της δικαιοσύνης γιατί σας έχει αφαιρεθεί δήθεν η κυδαιμονία των παιδιών. Επίσης σας λένε ότι ε, οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος Νεότητας ε, δεν ε, εκπροσωπούν κάποια επίσημη αρχή αλλά εκφράζουν μόνο την προσωπική τους εκτίμηση, άρα δεν μπορεί κανεί να του τριμώξει ούτε να προσφύγει εναντίον τους ενώπιον της δικαιοσύνης. Λέμε ότι πρέπει να ληφθεί ε, ε, υπόψη ο χρόνο. Δεκαετή είναι οι διαδικασίε ε, αυτές και επομένως ο ψυχικό μαρασμό των παιδιών βεβαίω δεν μπορεί να μετρηθεί και μπαίνει κανείς σε έναν φαύλο κύκλο ε, με άρνηση των δικαιωμάτων επίσκεψης, ε, με άρνηση όλων των αρχών ε, που διέπουν ακριβώς αυτή τη σχέση του γονιού με το παιδί. Εάν κανείς καταφέρει να κάνει μήνυση κατά του Ιδρύματος Νεότητος θα καταστραφεί οικονομικά. Κοιτάξτε, υπάρχουν όλο και περισσότερες ε, οικογένειες ε, οι οποίες ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του Ιδρύματος Νεότητας. και κανείς να ρίξει μια ματιά στο ίντερνετ. Και το πρόβλημα αυτό δεν θίγει, δεν πλήττει μονάχα τις οικογένειες, τους μεικτούς γάμους, αλλά και τους γερμανογερμανικούς γάμους. Μπορώ να σας αναφέρω περιπτώσεις, ας πούμε, όπου εκπρόσωπος του Ιδρύματος Νεότητος επισκέπτεται μια οικογένεια και λέει δεν μου αρέσουν τα έπιπλα, άρα αυτός είναι ο λόγος να σας εφερέσω τα παιδιά. Ε, στην αρχή του γεύματο αναρωτιόμαστε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν για όλα αυτά γιατί αυτά εμπίπτουν στο εθνικό δίκαιο. Εγώ προσωπικά ε, μπορώ να σας πω ότι είναι καθολικά ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουν ούτε σημαία Ιταλική ούτε Γαλλική, είναι καθολικά. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο σε 97% των περιπτώσεων αρνείται το να δώσει απόφαση δεν λέει ούτε ναι ούτε όχι. Λέει ότι δεν αποφασίζω. Διαπιστώνουμε επίσης ότι δεν υπάρχει σεβασμός του άρθρου 167 ε, της Βασικής Συνθήκης Λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διότι αρνείται το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της, ε, του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου λέγοντας ότι ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθούν, να συζητηθούν τα θέματα αυτά ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, κυρίως δεν ενώπιον του αερίου Πάγου. Καμία δυνατότητα προσφυγής δεν μπορεί να έχει κανείς, μια και δεν αναγνωρίζεται και το δικαίωμα έφεσης. Εγώ πιστεύω ότι, αν και είμαι Γερμανός, ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση κατά της Γερμανίας, παραβάση ε, ε, σε σχέση με τις συνθήκες λειτουργίας. Είμαι Γερμανός και ζητώ συγγνώμη από όλους τους ε, πάσχοντες γονείς. Υποφέρω και εγώ μαζί σας και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Άρης Χριστίδης. Θα μιλήσω γερμανικά παρότι είμαι Έλλην ε, πολίτης, όχι μεταναστής. Ναι, να πω καλησπέρα στα ελληνικά. Να ξεκινήσω, ε, επειδή δεν έχω προετοιμάσει, με το διαζύγιό μου το οποίο οριστικοποιήθηκε το 2005. Τα παιδιά μου εκείνη τη χρονιά ήταν 6 και 8 ετών και ο λόγος ήταν τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ε, η γυναίκα μου. Ήθελα να δημιουργήσω ένα νησί για τα παιδιά μου. Τα παιδιά ήρθαν σε μένα, δεν ήθελα να γυρίσουν. Εγώ όμως τα γύρισα στην πρώην γυναίκα μου. Θέλαμε να τα ε, μεγαλώσουμε μαζί αλλά όντας χωρισμένοι. Μετά το διαζύγιο λοιπόν άρχισαν και οι διακρίσεις εις βάρος μου. Ε, όταν ε, βγήκε το διαζύγιο ζούσα ήδη 35 χρόνια στη Γερμανία, είχα μια καθηγητική θέση και ζούσα ήδη στο Γκίσεν και ήμουνα και δημοτικός σύμβουλος. Και ε, είπα ότι θέλω να βλέπω τα παιδιά μου ε, το, το ίδιο συχνά όσο και η, γυναίκα, η πρώην γυναίκα μου. η δικαστής είπε ότι στη Γερμανία δεν ισχύει αυτό. Ε, ότι υπάρχει μια εναλλαγή, ε, ότι αυτό είναι το καθεστώς στη Γερμανία. Έτσι ξεκινήσαμε και η κατάσταση χειροτέρευε όλο και περισσότερο. Ένα χρόνο μετά μειώθηκε κατά 36% ο χρόνος ε, που είχα στη διάθεση μου με τα παιδιά για να μπορούν να παίζουν περισσότερο ποδόσφαιρο. Ε, μιλούσα διαρκώς με αυτό το Ίδρυμα Νεότητας και είχα πραγματικά την υποστήριξη δύο κυριών που ήταν υπεύθυνες ε, η μία κυρία αυτή μετατέθηκε, δεν ξέρω αν ήταν δυσμενή η μετάθεση της και η δεύτερη κάποια στιγμή μου έγραψε ότι μου απαγορεύτηκε να μιλά μαζί, της απαγορεύτηκε να μιλά μαζί μου. Το 2008 τα, τα παιδιά μου σταμάτησαν τα μαθήματα ελληνικών ε, με ευθύνη της γυναίκας μου ε, η οποία ελάμβανε συμβουλές να μην αφήνει τα παιδιά μαζί μου. Φυσικά προσέφυγα στο δικαστήριο και το, ε, το ανώτατο δικαστήριο της Φραγκφούρτης ε, επικύρωσε ότι τα παιδιά μου δεν πρέπει να μάθουν ελληνικά διότι ε, δεν δημιουργούσε ε, κάποιο πρόβλημα το γεγονός αυτό. Θα μπορούσα εγώ να τους διδάσκω ελληνικά και βεβαίως το να μην μιλούν ελληνικά δεν θα ήταν και πρόβλημα. Το πώς αποφασίστηκε όλο αυτό μπορώ να σας πω το εξής. μερικές εβδομάδες αργότερα ε, υπό τις φωνές της μάνας του ο μικρός γιος μου με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να επανέλθει, να επιστρέψει στα μαθήματα ελληνικών. Πράγματι πήγαινε τακτικά στα μαθήματα, έως το, στα μαθήματα ελληνικών, ε, ε, έως το καλοκαίρι του 2009, όπου πραγματικά τελείωσε όμως και αυτή η διαδικασία. το 2010 μετά δύο ε, ψυχολόγοι και ε, οι ε, ειδικοί ε, επιτετραμένοι ε, επιβεβαίωσαν ότι η, μητέρα κακοποιεί σεξουαλικά τα παιδιά της και το αποτέλεσμα ήταν ότι αρχικά έγινε διερεύνηση του, του σπιτιού μου. Ε, έγινε, υπήρξαν, εκφράστηκαν υποψίες μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαπιστώθηκε ποια είναι η, διεύθυνσή μου και αντιστοιχήθηκε σε μένα μια λάθος πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Ε, έγινε λοιπόν ύποπτος ότι εμπορευόμαστε ξένα παιδιά. Ζήτησα λοιπόν μια πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί ότι τα, παιδιά μου ήταν, ε, αντιμετώπιζαν προβλήματα και ότι έπρεπε να ε, σταλούν σε ψυχοθεραπεία. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή ζητήθηκε, ε, μου παρουσιάστηκε ένα τιμολόγιο άνω των 10.000 ευρώ, το οποίο και αποπληρώνω, αλλά παρόλα αυτά μου αφαιρέθηκε η κυδαιμονία. Και ο λόγος ήταν ότι είχα μαλώσει με τη μητέρα τους και ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να ζήσουν και με τους δυο μας. Στη συνέχεια ε, η μητέρα μετακόμισε στη Βρεύμη από το 2011. Ελπίζω τα παιδιά μου να ζουν. Τα, έχω δει μία φορά. Ε, μάλιστα τα, τα ίδια τα παιδιά μου είπαν ότι επιτέλους πρέπει να μιλάω γερμανικά μαζί τους και πλέον υπάρχει και ένας δικαστής ο οποίος το έχει πει αυτό ε, και επικύρωσε ότι για δύο χρόνια δεν θα πρέπει να ε, ε, δω τα παιδιά μου. Προσέφυγα λοιπόν και Ε, ο δικαστής μάλιστα είπε ότι αν κανείς γκουγκλάρει το όνομα Χριστίδης τότε καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Πράγματι, το 1999 είχα διαμαρτυρηθεί ενάντια στου βομβαρδισμού στη Γιουγκοσλαβία. Ο κύριος Ζολί. Με, με συγχωρείτε, είμαι τυφλός, δεν βλέπω, άρα δεν μπορώ να προετοιμάσω, δεν μπορούσα να προετοιμάσω λόγο. Δεν θα πω πολλά για αυτά που έγιναν. Έχει την αναφορά. Υπήρξαν διακρίσεις σε βάρος μου λόγω της ε, αδυναμίας μου, λόγω της αναπηρίας μου. Μου υπόθηκε ότι δεν μπορούσα να αναθρέψω τα παιδιά, τα παιδιά μου. Αυτό ισχύει μόνο εάν δεν είσαι Γερμανός, γιατί οι Γερμανοί με αναπηρίες, με ειδικές ανάγκες, μπορούν να αναθρέψουν παιδιά αλλά όχι. Έγινε μια ανώνυμη καταγγελία κατόπιν ότι ήθελα να απαγάγω τα παιδιά μου. Αλλά δεν ήταν ανώνυμη, ήταν γνωστό το όνομα. Η κυρία αυτή είπε ότι ίσως είχα πρόθεση να απαγάγω τα παιδιά μου. Από τότε δεν ξαναείδα την κόρη μου. Μετά είδα την κόρη μου ε, υπό επιτήρηση. Από το 2009 την έβλεπα Τρει ώρε κάθε τρει εβδομάδε Πήγαινα από τη Γαλλία στη Γερμανία για να δω τρει ώρε, μια φορά κάθε τρει εβδομάδε, Έκτοτε δεν ξέρω ακριβώ. εδώ και τρία χρόνια κάνω αυτά τα ταξίδια το Σάββατο 10 με 18 και την Κυριακή 10 με 18 χωρίς δυνατότητα στέγασης. Γιατί μπορεί ακόμη να είχα πρόθεση να την απαγάγω. Είμαι τυφλός, δεν μπορώ να αναθρέψω τα παιδιά μου, θα μπορούσα να τα απαγάγω, να κρυφτώ από την αστυνομία, να ζήσω παράνομα, να περάσω από φράγματα. Οι Γερμανοί θεωρούν ότι όλα αυτά είναι δυνατά για μένα. Τι έγινε μετά. Εδώ και αρκετά χρόνια κάνω αυτά τα μπρος πίσω, φυσικά μου κοστίζουν τρομερά, με κουράζουν. Είναι ψυχολογικό βάσανο. Το κάνω κάθε τρεις εβδομάδες με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας ε, τυφλός για να κάνει τέτοια ταξίδια. Η κόρη μου επειδή δεν κατάφεραν να με κάνουν να τη βλέπω μόνο σε ένα χώρο υποδοχής του Ιδρύματος για την Νεότητα, βρήκαν άλλο τρόπο, ούτως ώστε η κόρη μου να μην μιλάει παρά μόνο γερμανικά. Ήδη από τεσσάρων ετών άρχισε να μου λέει ότι δεν ε, μπορώ να μιλήσω παρά μόνο γερμανικά, δεν μπορώ να μιλήσω γαλλικά γιατί θα μου ε, δημιουργήσει πονοκέφαλο. Αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία λοιπόν ο γερμανικός πατριωτισμός. Ας έρθουμε τώρα στην παρούσα κατάσταση. Πολύ σύντομα αντιλήφθηκα ότι η πρώην σύντροφός μου που έφυγε γιατί δεν ήθελα να κάνουμε άλλο παιδό, παιδί, έφυγε με κάποιον άλλον. Αυτή λοιπόν να πήγα για την κόρη μου. Κατά τις διαδικασίες αντιλήφθηκα πολύ νωρίς ότι είμαι πισμένος ότι ήδη είχε χωρίσει με τον ε, επόμενο σύντροφό της. Σημαντική αλλαγή λοιπόν για τη ζωή Ενό μικρού κοριτσιού έπρεπε να ξεκινήσω μια νέα διαδικασία για να ζητήσω και πάλι την κυδαιμονία. Τότε υπήρξαν έμεσες αλλά σαφείς απειλέ του δικαστή που μου είπε θέλετε να συνεχίσετε τη διαδικασία, θέλετε πάλι να ζητήσετε την κυδαιμονία. Συνέχισα. Κατόπιν ήρθε κάποια επιμελήτρια, κάποια δικηγόρος η δικηγόρος ε, που ε, είναι αρμόδια για τα θέματα των συμφερών των παιδιών να με ρωτήσει μετά από ένα τέταρτο ήθελε ήδη να φύγει έπρεπε να την κρατήσω για να της εξηγήσω την άποψή μου και ήρθε χωρίς διερμηνέα δεν καταλάβαινα τι μου λέει τι έγινε μετά σύρθηκα ενώπιον των ε, δικαστηρίων δύο-τρεις ώρες ακρόαση έκαναν κάθε προσπάθεια να μου λένε ότι εγώ δημιουργούσα τα προβλήματα, ότι εγώ αποξένωνα το παιδί μου από μένα, ενώ οι προηγούμενοι δικαστές που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεση είχαν σαφώς αποφασίσει ότι η μητέρα είχε αποξενώσει το παιδί, αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να μείνει με το παιδί. Με κατηγόρησαν σε αυτή την νέα διαδικασία ότι εγώ αποξένω το παιδί μου από μένα. Ζήτησα να αλλάξει ο δικαστής, να εξαιρεθεί αυτός ο δικαστής και τι έγινε τότε. Αν ζητήσει την εξαίρεση ενό δικαστή, οι συνάδελφοί του, του ίδιου γραφείου αποφασίζουν εάν θα εξαιρεθεί ή όχι. Ζήτησαν λοιπόν από τον αντίδικο να απαντήσει εάν ο δικαστής ε, είχε μεροληπτήσει υπέρ κάποιας πλευράς. Ζητούν από τον αντίδικο να πει αν είναι αμερόληπτος ο δικαστής. Καταπληκτικό. Πρωτόγνωρο. Μου κόστησε και αυτό αρκετές εκατοντάδες ευρώ τι έγινε μετά. Η κυρία Πασολιέ με την οποία ζω εδώ και χρόνια να αναφέρω στην αναφορά μου ο πρώην σύντροφ κύριε σας παρακαλώ να τελειώνετε 30 δευτερόλεπτα ακόμη ο πατέρας λοιπόν ε, ο πατέρας των παιδιών της συντρόφου μου μου έκανε μήνυση για βιοπραγίες κατά των παιδιών και της συντρόφου μου. Έγινε ανάκριση, ερώτησαν τα, παιδιά, ρώτησαν όλο το περιβάλλον του πρώην συντρόφου τους για γεγονότα που είχαν συμβεί στη Γαλλία. Δεν ρώτησαν όμως ε, μάρτυρες στη Γαλλία. Και σήμερα επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα άλλο, βεβαίως ε, με απείλαξαν. Σήμερα λοιπόν καταδικάστηκα, έχω ήδη καταδικαστεί σε 80 μέρες φυλάκιση και 2.500 ευρώ πρόστιμο. Ε, περιμένουμε ακόμη την απόφαση, ε, γιατί έχω κάνει βέβαια έφεση, αλλά θα επικρέμαται. Και αν μια, μια μέρα αποφασίσουν να με καταδικάσουν γιατί τους ενοχλώ, τότε θα με καταδικάσουν. Ευχαριστώ κύριε Ζολίου. Έχει ζητήσει και κάποιος άλλος το λόγο νομίζω. Ε, κύριος ε, Πούτκιν. Πολύ σύντομα, αυτό το διοικητικό μέτρο το οποίο, ε, ε, το οποίο θεωρεί η Γερμανία ότι ε, χρησιμοποιεί ως μέτρο με νομική ισχύ έτσι ώστε να μπορεί να παίρνει χρήματα από, όλες τις, από τους ενδιαφερόμενους από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Χρησιμοποιείται και στην περίπτωση Τζιλμπέρτη και στην περίπτωση Πούτιν. Σε περίπτωση που ένα παιδί ε, απαχθεί προς τη Γερμανία, τη στιγμή που το παιδί, αυτό το απαχθέν ε, παρανόμος ε, παιδί πηγαίνει στην Γερμανία, ο γονιός αυτός, ο απαγωγέας, μπορεί να ε, πάει στο Ίδρυμα για την Νεότητα, να ζητήσει μια προκαταβολή χρημάτων και να τελειώσει το θέμα. Εδώ μιλάμε για μια απόφαση η οποία είναι διοικητική και όχι νομική. Είναι μια απόφαση όμως η οποία αντιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, και αντιτίθεται ε, σε όλες τις νομοθεσίες οι οποίες διέπουν τις μεθοριακές κινήσεις. Γιατί δίνονται χρήματα σε ένα είναι απαγωγέα Γερμανό. Βεβαίω αυτή είναι λέξη η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, την γερμανική πλευρά, ωστόσο αυτή είναι η αλήθεια. ενα ε, Γερμανός ε, ο οποίος έχει απαγάγει παράνομα και έχει πάρει παράνομα ένα παιδί στη Γερμανία από τη στιγμή που του δίνει χρήματα το Ίδρυμα για την Νεότητα σημαίνει ότι τον, του δίνει άφηση αμαρτίων και δεν τον θεωρεί πλέον εγκληματία και απαγωγέα. Ο, κύριος Ζολή. Ε, κοιτάξτε, πρέπει να ακούσουμε τώρα τους ευρωβουλευτές. Ναι, μονάχα ένα ερώτημα το οποίο δεν έθεσα προηγουμένως. Η αναφορά μου θεωρήθη παραδεκτή ε, και ε, ορίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική έρευνα. Αλλά δεν έχω όμως κανένα νέο επ' αυτού. Έχω... Τέσσερις βουλευτές έχουν τον λόγο. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα. Ξέρετε πρέπει να τελειώσουμε στις 6.30. Μπουρλά, Βίλαντ, Μπέρμαν και ο Ιραθαβαλέτια. Ο κύριος Μπουρλά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν ήθελα να πάρω μέσα στο λόγο, δεν πειράζει. Ήθελα να ζητήσω τους συναδέλφους, να αφήσω τους συναδέλφους να πάρουν το λόγο. Εν πάση Θεωρώ ότι από αυτά που ακούσαμε από τους αναφέροντες φαίνεται η έκταση του προβλήματος έναντι μιας μηχανής διοικητικής και δικαστικής που τους καταπνίγει και προσωπικά γιατί δεν έχουν ε, τα μέσα για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μηχανή ούτε οικονομικά ούτε στήριξη οικογενειακή, επαγγελματική και βλέπετε τι επίπτωση έχει αυτό σε κάθε επίπεδο. Αν θέλουμε να εξαγάγουμε πορίσματα από όλες αυτές τις τόσο κραυγαλαίες περιπτώσεις, δεν μπορούμε παρά να συγκινηθούμε γιατί έχουμε καρδιά ως Επιτροπή Αναφορών. Εμείς ε, προερχόμαστε από τους Ευρωπαίους πολίτες Πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε απαντήσεις ε, στις αναφορές που κρίθηκαν παραδεκτές. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε απαντήσεις. Επιπίων θεμάτων πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Είναι ότι υπάρχουν διακρίσεις σε σχέση με τα διοικητικά διαβήματα που πρέπει να κάνουν σε μια ξένη χώρα Ορισμένοι βέβαια μιλούν τη γλώσσα, αλλά όλοι αυτοί οι διοικητικοί μηχανισμοί είναι υπερβολικά περίπλοκοι, λαμβάνονται παράνομες αποφάσεις. Την παραμονή πολλές φορές ε, της ε, άφηξης του πατέρα για να ασκήσει το δικαίωμα επίσκεψης, λαμβάνεται απόφαση ότι δεν έχει πια δικαίωμα επίσκεψης και αν επιμείνει μπαίνει φυλακή υπάρχει άρνηση να σεβαστούν ε, αποφάσεις άλλων χωρών τα γερμανικά δικαστήρια γιατί σε μία περίπτωση που δεν ε, ομίλησε ο αφορόμενος υπήρχε μία απόφαση γαλλικού δικαστηρίου που αφισβητήθηκε από τις γερμανικές αρχές και αυτή την υπηρεσία νεότητας. Ή πρέπει να υπάρχει σύνδεση και μεσολαβητές μεταξύ των ε, δικαστηρίων και δικαστές ειδικευμένοι γιατί εκδίδουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης μόνο με ε, την υποψία ότι μπορεί να απαγάγει ένας γονιός το παιδί που παίρνει απλώς για διακοπές. Γιατί κάποιος που υποτίθεται δεν πληρώνει διατροφή, παρά το ότι έχει πληρώσει παραπάνω από ό,τι έπρεπε, γιατί να εκδίδεται και κατά του πολίτη αυτή, αυτού τέτοιο ένταλμα ασύλληψης και να φυλακίζεται. Υπάρχουν διαδικασίες και αστικού δικαίου που μπορούν να αξιοποιηθούν πριν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Όλη αυτή η διαδικασία είναι σαν από βιβλίο του Κάφκα. Κάναμε διερευνητική επιτροπή ε, επίσκεψη συγγνώμη, στο Βερολίνο, δεν βγάλαμε τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα πόρισμα και καμία βοήθεια από τις γερμανικές αρχές για τις προηγούμενες αλλά και για τις επόμενες αναφορές από αυτή τη διερευνητική αποστολή. Ίσως πρέπει λοιπόν να επιχειρήσουμε να τους ταράξουμε λιγάκι τους Γερμανούς φίλους μας να τους πούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας η συμπεριφορά σας μπορεί να θεωρηθεί μη βοήθεια σε άτομο κινδύνο μη βοήθεια σε πολίτη της Ευρώπης εν κινδύνο, σε παιδί εν κινδύνο, θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ανεξαρτήτως της υπηρεσίας νεότητας που να επιτρέπουν να αμφισβητηθεί η δράση της υπηρεσίας νεότητας, να αμφισβητηθούν οι αποφάσεις δικαιοσύνης, ούτω ώστε άτομα που δεν ελέγχονται να μην μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που καταστρέφουν τη ζωή ε, πολλών ατόμων της ίδιας οικογένειας. Τι θα γίνει. Είμαστε στο έτος ευρωπαϊκής ε, ηθαγένειας. Είμαστε ενώπιον των εκλογών. Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτές, αυτά τα μεγάλα ιδανικά ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα να αγαπάει κανείς ένα Γερμανό ή μια Γερμανίδα χωρίς να κινδυνεύει να χάσει τα παιδιά στο μέλλον. Θα ήθελα λοιπόν να παραμείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προειδοποίηση προς τη Γερμανία να αναλάβει τις ευθύνες της να υπάρξουν διαδικασίες για να βοηθήσουν αυτούς τους γονείς, αυτές οι οικογένειες για κατά τη γνώμη μου πρόκειται για περίπτωση μη βοήθειας ατόμων εν κινδύνου. Ο κύριος Βίλαντ. Δεν είχα ζητήσει το λόγο. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το ε, επίδομα θα ήθελα να ακούσω κάτι από την Κομισιόν διότι έχουμε να κάνουμε ε, με ένα νέο ζήτημα. Ε, θέλω να πω ξεκάθαρα ότι το αντικείμενο των αναφορών μπορεί, μπορούν να είναι μόνο εκείνα που αφορούν διασυνοριακά τους πολίτες της Ένωσης και αυτό διότι δεν είναι Γερμανοί πολίτες. αυτό είναι το, το, το, ο λόγος για τον οποίο οι αναφορές ε, ε, ε γίνονται αντικείμενο συζήτηση εδώ στην Επιτροπή. Το είχαμε συζητήσει και πριν από 5-6 χρόνια, ώστε σε αυτές τις περιπτώσεις να γίνονται παραδεκτές αυτές οι αναφορές. Το γεγονός ε, ότι ε, υπάρχουν και προβλήματα σε κάποια χώρα ή ότι ε, αποδεικνύονται αποφάσεις ως εσφαλμένες αντικειμενικά αυτό είναι αναμφισβήτητο. Σε μια μεγάλη χώρα βεβαίως αυτό συμβαίνει πιο συχνά από ότι σε μια μικρή. Εξαρτάται και από τον πληθυσμό. Η δικαιοσύνη δεν είναι τέλεια. Ωστόσο, αντικρούω ότι όλο αυτό είναι μεθοδευμένο. Σας άκουσα. Και δεν σας διέκοψα ούτε μία φορά. Παρακαλώ να μην το κάνετε ούτε εσείς. Διότι αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε να συζητάμε. Ε, κύριε ε, Μπουλάν, το χρονοδιάγραμμα που ε, αποφασίσαμε στο Βερολίνο ήταν πολύ στενό. Είχαμε μιλήσει με ε, Γερμανούς και Γάλλους δικαστές. Υπήρχε ένας Γάλλος δικαστής ο οποίος είπε ε, ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς κάνουν λάθος οι Γερμανοί δικαστές. Μάλιστα υπήρχε και η πρόταση να υπάρξει ε, επίσκεψη σε μια διαπραγμάτευση δικαστική. Εσείς φταίτε για το γεγονός ότι δεν έγινε τελικά αυτή η επίσκεψη και με εκπλήσει το γεγονός ότι εσείς χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα. Να το πω σαφώς οι περιπτώσεις παραβίασης ε, ε, της ε, πληρωμής διατροφής ε, δεν, έχει δεν έχουν σχέση με το, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η Χάρτα των ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεσμεύει τα κράτη-μέλη στο να εφαρμόζουν το, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο έδαφος τους. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει αυτή η Χάρτα και να δεσμεύει τα, όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ε, η τρέχουσα κατάσταση είναι αυτή ε, και ε, πρέπει να αναλαμβάνονται δράσεις όταν πράγματι έχουμε ευρωπαϊκές υποθέσεις αλλά η παραβίαση της πληρωμής των, της διατροφής δεν έχει καμία θέση εδώ και πρέπει να σας πω κύριε Μπουλόν ότι είναι κάπως περίεργα αυτά που μας είπατε το ότι πληρώθηκε περισσότερα χρήματα σε διατροφή. Ωστόσο δεν υπάρχει κανένας τρόπος αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν. Ούτε μπορεί κανείς αντλήπιτουμ να πει ότι τώρα δεν πληρώνω τίποτα γιατί δεν μου αρέσει το ένα ή το άλλο στοιχείο. Και στην Γαλλία φυσικά θα πάει κανείς φυλακή αν το κάνει αυτό. Από αυτή την άποψη είναι ε, εντελώς φυσιολογικό όταν υπάρχουν παραβιάσεις της πληρωμής διατροφής να υπάρχουν και επιπτώσεις. Ε, θέλω να εκφράσω το σεβασμό μου προς τους αναφέροντες που είπαν με, τόση, ε, με τόσο θάρρος ότι έχουν προβλήματα και με τον νόμο. Ωστόσο θέλω να ρωτήσω ρητά την κυρία Κολόμπο ε, που είπε ότι η δικαιοσύνη την χαρακτήρισε εγκληματία. Εγώ δεν το έκανε. Δεν το έκανα αυτό. Ε, το, να το πει Ποιο ε, δικαστής αυτό είναι ιδιαίτερο ε, σε αυτή την περίπτωση ε, αντιμετωπίζει κανείς κάθεξη ενός έτους τουλάχιστον εγώ δεν θα σας χαρακτηρίσω εγκληματία αλλά θέλω να σας ρωτήσω ρητός έχετε καταδικαστεί από δικαστήριο, από γερμανικό δικαστήριο, από ιταλικό δικαστήριο και ποια ακριβώς είναι η αξιόπινη πράξη και αν ε, καταδικαστήκατε και σε κάθερξη ή αν ε, είχε αναστολή η ποινή που σας επιβλήθηκε. Θα ήθελα να το μάθω αυτό. Πρέπει να απαντήσω. Ναι. Να, ναι, σας έκανα άμεσα την ερώτηση, αλλά απαντήστε. Ναι. Λοιπόν, απαντώ. Πρώτα απ' όλα, αποσαφήνισε ο Μιλών ότι είναι ε, η Δήμων για θέματα οικογενειακού δικαίου και εγώ γιατί στην Ιταλία οι εγκληματίες ε, τελειώνουν τις σπουδέ τους και γίνονται εμπειρογνώμονες. Σε πάση περιπτώσει εκρεμεί μια απόφαση ε, της εισαγγελία του Μιλάνο, όπου αναφέρεται μπορώ να σας δώσω και το χαρτί, ότι ο Γερμανός δικηγόρος του συζύγου μου πλαστογράφησε την ε, μετάφραση και βάσει αυτού του εγγράφου του ε, πλαστογραφημένου ε, υπάρχει απόφαση δικαστηρίου του Μιλάνου που έστειλε τα παιδιά μου στη Γερμανία. Ε, Quiero Τελειώσουν οι βουλευτές. Θα έχουν πολύ σύντομα το λόγο οι αναφέροντες. Κυρία Βέρμα. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά συμφωνώ με τον συνάδελφο Βίλαντ. Υπάρχει πρόβλημα όταν ε, συζητάμε αναφορές που ασχολούνται με θέματα διατροφής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι πρόβλημα εθνικού δικαίου, όχι ευρωπαϊκού δικαίου. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρος. Έχετε επανειλημμένα, επανειλημμένα διακόψει. Σας παρακαλώ. Νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα ε, άνετοι μέσα. σας. παρακαλώ να μην, να μην ε, διακόψετε άλλη φορά την κυρία Μπέρμαν. Ευχαριστώ πολύ. Σέβομαι τους αναφέροντες που μας παρουσίασαν τα προβλήματά τους, αλλά εμείς ως βουλευτές έχουμε καθήκον να συμβουλεύουμε τους αναφέροντες, να τους ε, πλαισιώνουμε για το εάν πρόκειται για παραβίαση ευρωπαϊκού δικαίου ή όχι. Υπάρχουν βέβαια διοικητικά προβλήματα, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα διάκρισης. Ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας του Βερολίνου. Τα ξέρω τα θέματα αυτά. Και νομίζω ότι στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούλιο ή το φθινόπωρο της Επιτροπής μας θα πρέπει να συζητήσουμε και ως συντονιστές το θέμα αυτό. Κύριε Μπουρλά, ένα θέλω να σας πω και εγώ γνωρίζω ότι αντίστροφα υπάρχουν και Γερμανοί γονείς ε, των οποίων τα παιδιά απέκτησαν στη Γαλλία και δεν επεστράφησαν με την απλή εξήγηση ότι θα γερμανίζονταν υπερβολικά. Εγώ δεν πρόκειται τώρα να πω ότι είναι σωστό ή όχι και να πάρω αποφάσεις θα ήθελα να το παρατηρήσω αυτό, ότι εμείς ως βουλευτές πρέπει να ασχολούμεθα μόνο με τα θέματα που πραγματικά αφορούν ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο και το παραβιάζουν. Και για τέτοια θέματα πάντα είμαι πρόθυμη να συζητήσω. Αυτό ήθελα να πω προς τους αναφέροντες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βεντάνη. Ο κύριος Ιρεθαβαλβέτια. Αυτό που ακούσαμε εδώ μου θυμίζει αυτά που ακούσαμε πριν από δύο εβδομάδε για παρόμοιε περιπτώσει στη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε πιστεύω. Δεν ξέρω εάν παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο, γιατί είναι γενικότερο πρόβλημα. Πρέπει να μας απαντήσει η Κομισιόν για να δει εάν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Θέλω να, παραμείνει ανοιχτή, να παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές και αυτό που είναι σοβαρό είναι ότι είναι σοβαρό ε, αυτό που συμβαίνει και στη Μεγάλη Βρετανία ότι απαγορεύουν σε γονείς να βλέπουν τα παιδιά τους. Πρόκειται λοιπόν για διάφορες περιπτώσεις είναι τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των γονέων, τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή δεν ξέρω αν θα ζητηθεί στην επόμενη θητεία γιατί εγώ δεν θα είμαι αλλά θεωρώ ότι επίσης πρέπει να πούμε στην Κομισιόν να ασχοληθεί με το θέμα αυτό να μελετήσει την υποβολή νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφεύγονται τέτοια θέματα μεταξύ χωρών της Ένωσης Έχουμε θέματα τέτοιου τύπου βρετανικά, δανέζικα, ε, γερμανικά και θα υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ένωσης. Τέτοιου τύπου προβλήματα πρέπει να επιληθούν επαρκώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Ραθαβαλβέτια. Για να δούμε τώρα. Μισό λεπτό. Έχετε υποβάλει έκθεση. Κοιτάξτε, όχι, δεν γίνεται έτσι. Ποιο θέλει να μιλήσει από του αναφέροντε για να απαντήσει σε ερωτήσει. Ωραία. Δύο λεπτά ο καθένα Και στον κύριο. Δύο λεπτά παρακαλώ. Παρακαλώ αρχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ δεν ήρθαμε να συζητήσουμε προβλήματα σχετικά με τη διατροφή. Εγώ ήρθα εδώ ε, γιατί ε, είπα ότι ε, παρεπιπτόντως τα, παιδιά χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να στέλνονται χρήματα στη Γερμανία. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αρνούνται στα παιδιά τον ένα γονιό τους, μητέρα ή πατέρα, με την δικαιολογία μόνο και μόνο γιατί δεν είναι Γερμανός. Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, ε, άνθρωποι, όχι μονάχα Γερμανοί, οι οποίοι γνωρίζουν καλά το γερμανικό ε, δίκτυο. Πήγατε στην Γερμανία, συζητήσατε με την Γερμανίδα δικαστή για τον αστικό κώδικα της Γερμανίας, αλλά ε, αποσιωπούν τον κοινωνικό ε, κώδικα ο οποίος διευθετεί όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την νεότητα μεταξύ ε, αυτών και την λειτουργία του Ιδρύματος για την νεότητα και αυτό δεν είναι σωστό. Όταν μιλάμε για δικαιώματα πρέπει να μιλήσουμε για ευρωπαϊκά δικαιώματα αλλά στη Γερμανία υπάρχουν δικαστήρια τα οποία μπορούν να στα οποία μπορούν να προσφύγουν οι γονείς έτσι ώστε να αποκτήσουν την κυδαιμονία του παιδιού ε, και η κυδαιμονία δίνεται βάση του γερμανικού νόμου μονάχα εάν το δικαστήριο το ίδιο θεωρήσει ότι μπορεί το παιδί να μεγαλώσει με τις σωστές προϋποθέσεις και όρους. Αυτό αν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο τι να σας πω. Πρέπει να πω ότι είχα μεγαλύτερες προσδοκίες από τους Γερμανούς Ευρωβουλευτές. Αυτό που άκουσα ε, το τι ε, άκουσα το τι δεν πρέπει να συζητείτε εδώ και ότι υπάρχουν και αδικίες και σε άλλες χώρες. Ε, εγώ ως Έλληνας λοιπόν τώρα μπορώ να αισθάνομαι καλά ότι όσο μένω στη Γερμανία και πληρώνω δεν θα υφίσταμαι τις αδικίες του δανέζικου συστήματος. Δεν είναι αλήθεια. Είναι λάθος να προσπαθείτε να μας πείσετε ότι δεν υπάρχει σύστημα. Πριν είπα ότι πλήρα, πλήρωσα 10.000 ευρώ για μια πραγματογνωμοσύνη και σας είπα ότι η πραγματογνωμοσύνη αυτή υπάρχει ήδη. Και μάλιστα έλεγε αυτή η πραγματογνωμοσύνη ότι είμαι παρανοϊκός και μάλιστα ε, ε, χρησιμοποιήθηκε για να απολυθώ ως δημόσιος υπάλληλος το, η πραγματογνωμοσύνη αυτή αποσύρθηκε, παρόλα αυτά όμως πρέπει να την πληρώσω. Στην Έση και στη Βρέμη έχω, ε, ε, έχω ε, λάβει επιβεβαιώσεις ότι τα παιδιά μου δεν μαθαίνουν ελληνικά, όχι για κάποια, με κάποια αιτιολόγηση, όχι δεν μαθαίνουν ε, ελληνικά. Ούτε τους ανανεώνονται τα διαβατήρια, διότι η μητέρα ε, ασκεί τα δικαιώματά της και ε, μπορεί να μην αιτηθεί ελληνικό διαβατήριο. Αλλά το, το γερμανικό διαβατήριο δίνεται στα παιδιά μου και χωρίς τη δική μου συνένεση. Είναι σύστημα, δεν είναι μονομενή περίπτωση. η η, η, απέτηση να, να μιλώ με τα παιδιά μου γερμανικά μου απευθύνθηκε στην Έση και στη Βρέμη, αλλά εγώ είμαι Έλληνας. Όλοι οι φίλοι μου είναι στην, στην Ελλάδα. Εγώ θέλω τα παιδιά μου που είναι πλέον 14 και 16 ετών να μιλούν ελληνικά. Και τέλος παρακάλεσα τουλάχιστον να καταγραφεί ότι τα παιδιά μου δεν κακοποιήθηκαν αλλά δεν, δεν, δεν υπήρξε καμία ερώτηση προς την ε, πρώην γυναίκα μου. Αυτό είναι, είναι συστηματική μέθοδος που ακολουθείται. Αυτό θέλω να πω. Ε, Πολύ σύντομα. Ε, συνεχώς ακούμε ε, παραπομπές στην εθνική νομοθεσία και ε, ρωτώ σοβαρά για ποιο λόγο η Γερμανία υπογράφει ε, διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλα θέματα όταν δεν έχει την πρόθεση να τηρεί τις συμβάσεις αυτές. Η Γερμανία υποχρεούται ε, να διασφαλίζει για παράδειγμα ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ε, βλέπουν και τους δύο γονείς τους και μια εξαίρεση μπορεί πραγματικά να υπάρξει μόνο σε πολύ εξαιρετικέ περιπτώσει όταν τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο. Και αν δείτε την πρακτική στη Γερμανία, είναι πραγματικά μια παραβίαση καραμπινάτη της, των ε, πρακτικών, των, ε, των διεθνών συμβάσεων. Για ποιο λόγο η Γερμανία λοιπόν υπογράφει τέτοιου είδου συμβάσει και για ποιο λόγο όλη αυτή η στάση γίνεται αποδεκτή. Also in Punkt, da bin ich jetzt voll und ganz bei Ihnen. Kinder, egal. Συμφωνώ. Τα παιδιά, όπου και αν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, έχουν δικαίωμα να ε, βλέπουν και τους δύο γονείς τους. Δεν, το συζητούμε αυτό. Και από αυτή την άποψη να εκφράσουμε την υποστήριξή μας στους αναφέροντες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε διεξοδικότερα. Ε, τα δικαιώματα των παιδιών πρέπει να τηρούνται και να ελέγχεται η τήρησή τους. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα γιατί ήδη οι διερμηνείς μας έχουν παραχωρήσει περισσότερο χρόνο από τον συνηθισμένο χρόνο εργασίας τους, ο οποίος έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Είμαστε απολύτως στη διάθεσή σας. Μπορούμε να συνεχίσουμε στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Δεν είναι πρόβλημα για μας. Ε, δεν ξέρω πώς θέλετε να συνεχίσουμε. Δύο, δύο λόγια να πω, δύο λόγια να πω στα Ιταλικά. Ε, θα, ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παραμένουν ανοιχτές αυτές ε, οι αναφορές έστω και ε, χωρίς να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μακροζωία εύχομαι στην Ευρώπη, όχι όμως στην Ευρώπη που είδα σήμερα εδώ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση και σε τούτες που παρουσιάστηκαν και σε όλες τις σχετικές αναφορές. Να πω κι εγώ ένα πραγματάκι Δύο λόγια με μικρόφωνο παρακαλούμε, δεν ακούν οι διερμηνείς. Το μικρόφωνο σας, το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ήθελα απλώς ε, να πω ότι είναι προφανές ε, ότι χρειαζόμαστε, πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Πρέπει να απαντήσω. Αν μου πείτε το όνομά σας, δεν το ξέρω δυστυχώς δεν με καλέσατε. Τουλάχιστον δεν έχω μάθει για κάποια πρόσκληση που έλαβα ότι θέλετε να μιλήσουμε. Φυσικά και θα μιλήσω μαζί σας. Κανένα πρόβλημα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ειδικά, ειδικά όταν ε, το θέμα αφορά παιδιά μπορεί να έρθει σε μένα και θα τον ακούσω. Και το επόμενο βήμα που ακολουθώ συνήθως είναι ότι θα κοιτάω τα έγγραφά σας και προσπαθώ να διαπιστώσω που ε, ε, υπήρξε παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικός όταν με κατηγορείτε. Όχι. Πρέπει να τελειώσουμε γιατί οι διερμηνείς πρέπει να φύγουν. Ε, Ρακέλ, σε παρακαλώ. Όταν λέει ότι πρέπει να μείνω εδώ, συγγνώμη, αλλά θα αμυνθώ. Διότι ειδικά όσον αφορά τα παιδιά, εγώ πάντα μένω. Συγγνώμη, έχω καθυστερήσει, πρέπει να φύγω. Έχω συνάντηση στις 7. Δεν μπορώ δυστυχώς να κάνω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να μείνω άλλο. Έχει περάσει ο χρόνος και επιμένω. Ευχαριστώ όλους που παρενέβησαν. Πρέπει να κλείσει το θέμα. Η αναφορά βεβαίως παραμένει ανοιχτή. Πολύ σύντομα. Σας παρακαλώ. Ήθελα να απαντήσω στους αδέρφους μου να πω στην κυρία Βέρμαν ότι υπήρξαν περιπτώσεις και στην Αυστρία και αν μιλάμε για την υπηρεσία νεότητας είναι γιατί έχουμε εκατοντάδες περιπτώσεις. Θέλω να πω στον κύριο Βίλαντ που δεν είναι παρόν που έφυγε με θάρρος πριν λήξει συζήτηση ότι συμφωνώ όταν λέει ότι δεν είναι η διατροφή θέμα αλλά όταν πληρώνει τη διατροφή και γι' αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκού και γίνεται μετά ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ε, αυτό είναι πρόβλημα. Ευχαριστώ και περιμένουμε την άποψη της Επιτροπής. Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και δεν είμαι εγώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ε, είμαι τόσο απογοητευμένος όσο και εσείς για την απουσία της, θα μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι διαμαρτυρίε σας, θα καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, στείλει και να σας στείλει στον καθένα σας η γραμματεία μας θα φροντίσει να λάβετε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίσης θα απευθυνθούμε άλλη μια φορά στις γερμανικές αρχές θα τις καλέσουμε να λύσουν το πρόβλημα θα ε, μεταβιβάσουμε όλες σας τις διαμαρτυρίες και τα νέα επιχειρήματα θα στείλουμε και τα νέα επιχειρήματά σας θα απαιτήσουμε μία απάντηση και ελπίζω να μην ε, χρειαστεί να καθυστερήσουμε πολύ ακόμη να υπάρξει σύντομα απαντήσεις η θητεία μας ε, λίγη στις 25 Μαΐου αλλά στην επόμενη θητεία όποιοι και να είναι θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα και ζητά από τη γραμματεία να του το πει. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Λίγη συνεδρίαση. Λίγη συνεδρίαση. Α, ναι. Δύο θέματα του Β. Το, το 1200 και το 1300, 1248 και το 1300, αν δεν υπάρχουν σχόλια. Α, και ένα τρίτο. Από τους πράσινους για την Παρθελώνα, η 1364 να μείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Λίγη τα... Ωραιότατα. What was that? Είχαμε μια